της ημερήσιας διάταξης, εάν συμφωνείτε. Εάν συμφωνείτε, εγκρίνετε. Όσοι ήθιστε, η συνεδρίαση αυτή θα αναμεταδίδεται στο ε, διαδίκτυο. Έχουμε 23 γλώσσες για τη σημερινή συνεδρίαση ε, στην ε, διερμηνία. Πρώτο σημείο, λοιπόν, έχουμε στην ημερήσια διάταξη την ψηφοφορία. Σύμφωνα με την ε, ωραία παράδοση που έχει θεσπίσει ο πρόεδρος Μπούζεκ, θα κάνουμε έναν έλεγχο. Ας κάνουμε λοιπόν έναν έλεγχο για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Σας αρέσει η Επιτροπή Ήτρε, λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Α, η κάρτα σας δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Αυτό ίσως γιατί μπορεί να είναι η παλαιά, γιατί βλέπω πως είναι διαφορετικό χρώμα. Χρειάζεται να την ανανεώσετε. Ίσως μπορείτε να μας ε, να δείξετε πώς ψηφίζετε. Για να μετρήσουμε την ψήφο σας. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν για τις ε, τροπολογίες για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης 2020. Όλες οι κατηγορίες, η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει on block για να επαναφέρουμε τις τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της ε, ψηφοφορίας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα Ψηφίζουμε για τις τροπολογίες μία-μία. 50-65. Ήτρε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 56 και 83. Ε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 51-68 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση σας σοσιαλιστές είστε υπέρ για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 51-68 51-68 ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 50-49. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-50. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-65. 67. Ποιοι είναι υπέρ κατά Αποχές, έλεγχος 5167. 51-67. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 51-65. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50-51, υπέρ, κατά αποχές 5084. 50-84 ε, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-91 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος 50-91. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Πενήντα εξήντα και πενήντα ενενήντα τρία. Ποιοι είναι υπέρ. Πενήντα και πενήντα ενενήντα τρία. Ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Πενήντα Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 50-47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-98 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5103. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5092. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5095. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5127. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5128. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 53 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος για την 50 53 Πέρας, εγκρίνεται.

50-13 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 51-05 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50-14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50-85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-06 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος 5106 τέλος απορρίπτεται 5071 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5016 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5072 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5017 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5073 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5018 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5086 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5087 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5019 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5096 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51-11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57-74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51-12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54, 50-54 υπέρ, κατά απόχέ εγκρινεται εγκρίνεται. 51-13, α, όχι αυτή είχε καταπέσει. 50-78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 51-14 υπέρ, απόχέ. αποχές απορρίπτεται. 50-75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50-46 υπέρ κατά αποχές δεν είδα πολύ καλά τα χέρια σας 50-46 ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Πενήντα εβδομήντα εννέα. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-89 και 51-30 από κοινού ποιοι υπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50-80 και 51-31 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται 50-24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά. 51-15 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, σοσιαλιστές ε, έχουμε μία παραπανήσια ψήφο. So someone has to redraw the card. Κάποιος λοιπόν πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα του. Α, τώρα είναι σωστά, εντάξει. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50-99. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτή έχει καταπέσει. 50-56. Υπέρ. Κατά. Σοσιαλιστές είστε υπέρ. Μάλιστα. Εγκρίνεται. 50-57. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5036 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-41 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 51-42 υπέρ 51-42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51-77 υπέρ, κατά, έλεγχος ηλεκτρονικά. 51-57. Τέλος και γκρίνεται. 51-78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51-53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51-73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50-58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 α, όχι 51-20 και 51-56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50-90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-81, 51-47, 51-80 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 50-82 Α, που είναι ταυτόσημη 51-48 και 51-21. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 51-49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-50 υπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51-51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50-61 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-01 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. 5101 άρχεται. Η πράσινη έχετε μία παραπανήσια. Παρακαλώ κάποιος να αφαιρέσει την κάρτα του από τους πράσινους. Τώρα είναι εντάξει. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε 50, 62 και 51, 23. Περ, Πάλι δεν μπορώ να μετρήσω. Ε, ας ελέγξουμε. 50, 62 και 51, 22. ψηφίζουμε. Τέλος. Έγκρινεται. Συγγνώμη, δεν είδα τα, τα χέρια σας. 50-63, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-25. Τι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελικό σχέδιο για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. 51-26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51-63 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51-58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50-64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51-60 υπέρ κατά αποχές σοσιαλιστές είστε υπέρ ή κατά Πενήντα ένα. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51-79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51-82 ε, υπέρ κατά οι σοσιαλιστές τι κάνετε εγκρίνεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ποια ήταν μάλιστα να ελέγξουμε Τώρα το ΕΛΚΑ έχει μία παραπάνω ψήφο. Και απορρίπτεται. 50-77. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51-55. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Και τέλος. Δεν πάμε στο επόμενο. 5146 λοιπόν, 51-46. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51-56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 51-74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51-76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και νομίζω πως τελειώσαμε οπότε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες Τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη που είναι το 5. Πρόκειται για την ε, παρουσίαση μελέτης από ε, το θεματικό τμήμα πολιτικής Α. Πρόκειται για την ανάλυση της ανάπτυξης του 5G. you want to take your seats. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αν πάρετε τις θέσεις σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μόλις καθίσετε. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον δόκτωρα Colin Blackman και τον κύριο Simon Forge, συγγραφείς της έρευνας αυτής που προετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολιτικών ε, κατόπιν ε, αίτησης της Επιτροπής Ήτρε, της Επιτροπής μας. Ο κύριος ο Dr. Colin Blackman είναι διευθυντής του Comfort Associates με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας ως συντάκτης και σύμβουλος πολιτικών και κανονισμού σε αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή οικονομία. Υπήρξε συντάκτης ε, πολιτικών τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής πολιτικής κανονισμού και διακυβέρνησης, καθώς επίσης και Senior Research Fellow του CEPS, όπου και διεύθυνε το ψηφιακό φόρουμ. Ο κ. Simon Forge έχει επίσης περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία στην βιομηχανία της επικοινωνίας, κυρίως στην Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Είναι διευθυντής του SCF Associates Ltd, όπου ε, ε... όπου ειδικεύεται στις οικονομικές επιπτώσεις. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι Chartered Engineer. Η ανάλυση αυτή που θα μας παρουσιάσουν σήμερα εξετάζει σε βάθος τη συγκριτική ανάλυση της ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες ηγετικές οικονομίες όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η ανάλυση αυτή καθώς η τεχνολογία 5G σιγά σιγά αναπτύσσεται, παρόλο που τα στάνταρτ δεν είναι ακόμη οριοθετημένα και το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί δεν είναι ακόμη βέβαιο. Σήμερα λοιπόν στην παρουσίασή μας θα δώσω το λόγο στους δύο προσκεκλημένου μας και στη συνέχεια θα έχουμε ένα κύκλο διαβουλεύσεων. Στο τέλος βεβαίως θα έχουμε ε, Συζητήσει και σχόλια από τους δύο επιρογνώμονες. Να ξεκινήσουμε τώρα από τον κύριο Μπλάκμαν. Έχετε το λόγο κύριε Μπλάκμαν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Λέγομαι Κόλεν Μπλάκμαν και εδώ είναι ο συναδελφό μου Σάιμον Φόρτζ. Η ιστορία τώρα σε σχέση με την τεχνολογία 5G είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την σύντομη παρουσίαση που θα κάνουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα σας παρουσιάσουμε σύντομα λίγο το background σε ό,τι αφορά την βιομηχανία των ε, κινητών τηλεφώνων. Θα σας παρουσιάσουμε μια περίληψη των εκτιμήσεών μας σε σχέση με το πώς συγκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες ηγετικές οικονομίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ασιατικές χώρες, στην Κίνα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και θα σας προτείνουμε και τις συστάσεις μας σε πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε καλύτερα την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G τα επόμενα επόμενα χρόνια. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν σκεπτόμενοι την ε, βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας πριν την τεχνολογία 5G, τα τελευταία 30 με 40 χρόνια, νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει μια κάπως σταθερή εικόνα για παράδειγμα, ο αριθμός των ε, φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων έχει αυξομοιωθεί, αλλά όχι ιδιαίτερα. Βλέπουμε τον ίδιο εξοπλισμό, βλέπουμε τους ίδιους προμηθευτές στοιχείων, τα ονόματα που και που αλλάζουν, αλλά επί της ουσίας η κατάσταση παραμένει σταθερή. Βλέπουμε επίσης ο βαθμός κάθε της ενσωμάτωσης μεταξύ υπηρεσιών και υποδομής είναι επίσης κάτι που δεν έχει αλλάξει. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι μια σχετικά σταθερή εικόνα που έχει επιβιώσει την μετάβαση τεσσάρων γενεών τεχνολογίας από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Τώρα όμως πιστεύω ότι με την τεχνολογία 5G βλέπουμε τη δυνατότητα ε, μιας πολύ πιο έντονης κατάστασης στην ε, βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας. Και επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Σάιμον τώρα για να σας εξηγήσει γιατί. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, λέει ο κύριος Φόρτς. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε είναι τη βιομηχανία τεχνολογίας 5G και την προσέγγιση marketing, γιατί υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα marketing. Και πιστεύω ότι τα βασικά σημεία που είναι πολύ σημαντικά είναι ότι όλη αυτή η κούρσα της τεχνολογίας 5G race, 5G race όπως συχνά την αποκαλούν στον τύπο, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το κέρδος έχει να κάνει με την ανανέωση μιας κάπως λιμνάζουσας βιομηχανίας. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας, α, έχει πέσει η αξία τους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες αγοράς, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό κέρδος. Κανένας δεν έχει χρεοκοπήσει. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι υπάρχει μια έντονη πίεση από τους προμηθευτές. Αυτό που βλέπουμε είναι η όφηση να δίνεται από τους προμηθευτές, όχι από τον τομέα της ζήτησης. Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών που έχω δουλέψει για, όλη την, για το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου είναι διάσημη για να στηρίζει κάποια άλογα που είναι γκαραντή θα λέγαμε ε, και κάποια που ενδεχομένως και να αποτύχουν η ε, βιομηχανία έχει ένα ιστορικό όπου έχει στηρίξει τεχνολογίες που δεν ε, πηγαίνουν πουθενά. Σε ό,τι αφορά τώρα την κούρσα α, της τεχνολογίας 5G θα πρέπει να βασιστεί στις κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι προωθείται από τη βιομηχανική πολιτική μεταξύ των ε, μεγάλων κρατών προμηθευτών. Βλέπουμε αυτή την τεχνολογία 5G ε, μέσω ενός μακροοικονομικού φακού. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα είναι μια οικονομική κούρσα σε γενικές γραμμές η, κινητή, η τεχνολογία κινητής τηλεφωνία ήταν πάντα για τα χρήματα. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση αυτή τη στιγμή παγκοσμίω σε αφορά την κινητή τηλεφωνία. Αν ρίξουμε μια ματιά από πλευράς προμηθευτών στοιχείων, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η βιομηχανία πούλησε την ε, τεχνολογία 4G, LTE, Long Term Evolution, ε, πούλησαν και το LTEA, την Advanced μορφή της τεχνολογίας αυτής, πήραν τα χρήματα, τα ξόδεψαν. Τώρα λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμός, κυρίως από την Κίνα, από την εταιρεία Huawei, η οποία προτείνει αρκετές πολύ φτηνές συμφωνίες. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το δεδομένο αυτό αλλάζει τη βασική εξίσωση σε ό,τι αφορά την ε, βιομηχανία προμηθευτών της κινητής τηλεφωνίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να ταρακουνήσουμε την αγορά. Πρέπει να τους πουλήσουμε αυτήν τη νέα τεχνολογία. Και εδώ μπαίνει και η τεχνολογία 5G. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι η σωστή στιγμή για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων, τους MNOs. Δεν υπάρχουν επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζες και σας το λέω γιατί εγώ εργάζομαι στις τράπεζες και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σημαντική για την σωστή εγκατάσταση, τη γρήγορη εγκατάσταση, τη χρηματοδότηση. Οι τράπεζες δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν κατά πόσο είναι μια ασφαλής επένδυση η τεχνολογία 5G. Οι επενδυτές, εκτός ε, των ε, τραπεζικών κοινοτήτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως οι φορείς να απευθυνθούν, δεν μπορούν να καταλάβουν κατά πόσο υπάρχει εμπορική αξία στην τεχνολογία 5G. Οι φορείς ε, τώρα της κινητής τηλεφωνίας βλέπουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το λεγόμενο διαδίκτυο των πραγμάτων. Το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει να κάνει με την ε, διαχείριση μεγάλων δικτύων, ε, την ένωση εννέα διαφόρων τομέων. Αλλά όταν ρώτησαν κατά πόσο θέλουν να αγοράσουν ε, την τεχνολογία 5G, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι οι απαντήσεις που είχαμε από τους ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένους προμηθευτές είναι ότι για τους τομείς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή η τεχνολογία 5G, ο τομέας της υγείας, ο τομέας των τροφίμων. Αυτό που λένε είναι ότι ήδη έχουμε πολύ φτηνά τοπικά δίκτυα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι παραπάνω θα μας δώσει η τεχνολογία 5G. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να κοστίσει πολύ παραπάνω. Οι φορείς λοιπόν εκμετάλλευσης κινητού δικτύου θα ήθελα να έχουν αυτή την κάθετη συγκέντρωση στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως ε, τεράστια εμπόδια που θα πρέπει να υπερκαμφθούν. Υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης των δικτύων και η μεγαλύτερη φορεί εκμετάλλευση κινητής δικτύας θα χρειάζονταν νέες δεξιότητε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το μοντέλο. Οι προμηθευτές λοιπόν θέλουν να ταρακινήσουν την αγορά. Παρ' όλα αυτά, τόσο οι φορείς όσο και οι προμηθευτές δεν έχουν χρήματα για να επενδύσουν σε αυτήν την καινούρια γενιά τεχνολογίας. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα απευθυνθούν στις κυβερνήσεις γιατί δεν μπορούν να βρουν επενδυτές. Δυστυχώς όμως έχουμε εδώ μια κατάσταση κάπως σαν τα ρούχα του αυτοκράτορα θα λέγαμε. όσο πιο μεγάλη είναι η γενική άγνοια, τόσο περισσότερο λιμνάζει η εξαιρετική αυτή προσφορά. Και βεβαίως οι κυβερνήσεις πέφτουν σε αυτήν την παγίδα. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία αναφέρεται σε ένα ψηφιακό, την βλέπουμε σε ψηφιακά κράτη. Και υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που το παίρνουν πολύ σοβαρά. Καταλαβαίνουν ότι αυτή η τεχνολογία βρίσκεται εκεί σε ορισμένα κράτη για να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές. Το εξετάζουν. Λοιπόν, σε σχέση με άλλες ε, τεχνολογίες που θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τεχνολογία 5G δεν θα αντικαταστήσει την τεχνολογία LTE και LTEA. Είναι μια τεράστια επέκταση. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί γρήγορα. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί σε 10 με 15 χρόνια. Τα φάσματα συχνοτήτων είναι πολύ καινούρια. Είμαστε εδώ σήμερα και μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσω συστημάτων που δημιουργήθηκαν πολλά χρόνια πριν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι κάτι που χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι στην κινητή τηλεφωνία τόσο όσο εξετάζουμε σήμερα. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την εξάπλωση Ενέργε κεραίες, massive μήμο. Είναι σαν να μιλάει κανείς σε πάρα πολλού ανθρώπου το ίδιο ε, την ίδια στιγμή, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Η πυκνότητα των δικτύων μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Οι προηγούμενες γενιές τεχνολογίες, δούλεψα πολύ για την τεχνολογία 3G, χρειάστηκε 5 με 7 χρόνια για να υλοποιηθεί. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Ιδίω οι Κινέζοι ε, ξεκίνησαν τις ε, τεχνικές δοκιμές τους από το 2015 και έχουν ως στόχο το 2030 για να μπορέσει να εγκατασταθεί η τεχνολογία. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν δύο πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα που συζητάμε σε ό,τι αφορά την τεχνολογία 5G. Πρώτα απ' όλα είναι τα δίκτυα 5G ως αντικατάσταση της τεχνολογίας που έχουμε τώρα. Αυτό είναι ένα απλό μοντέλο που μπορούμε να το δούμε, είναι απτό. Κατά πόσο οι καταναλωτές ε, θα το θέλουν και κατά πόσο θα δούνε και θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτό το πιο γρήγορο δίκτυο ε, αυτή είναι μια άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιεί πολύ πιο υψηλές συχνότητε. χρησιμοποιεί πολύ πιο πυκνά δίκτυα και ίσως εκατό φορές περισσότερες κεραίες, περισσότερες σταθμούς βάσης. Το άλλο μοντέλο που ανέφερα και πριν είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και υπάρχουν και πάρα πολλοί τομείς που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ε, συμπεριλαμβανομένης και της ρομποτικής. Αυτό θα δούμε όμως πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Ποιοι είναι λοιπόν οι παγκόσμιοι υπέκτες ε, αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι θέσεις τους. Και εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό ήταν και το θέμα της εργασίας μας. Τι είναι ακριβώς αυτή η κούρσα για την τεχνολογία 5G. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε διαφορετικές χώρες. Από τη μία έχουμε αυτούς που παράγουν, που ε, προσπαθούν να βγάλουν χρήματα παγκοσμίω από αυτή την τεχνολογία. Απ' την άλλη, έχουμε του καταναλωτέ που θα αγοράσουν αυτή την τεχνολογία και μετά έχουμε τα κράτη που είναι τόσο παραγωγή όσο και καταναλωτέ. Η Κίνα ανήκει και στι δύο αυτέ κατηγορίε, η Ιαπωνία το ίδιο, τόσο παραγωγή όσο και καταναλωτέ. Η Νότια Κορία είναι κυρίω παραγωγό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αν ε, κοιτάξετε αυτέ τι τρει χώρε, Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορία τα μέσα δόθηκαν στους τρεις βασικούς πάροχους. Στην Κίνα συγκεκριμένα δόθηκε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει ένα δίκτυο e-commerce. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ηγούνται και τόσο πολύ τη κούρσα αυτή, δεν είναι και τόσο πολύ μπροστά μα. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μπροστά σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση. Βλέπουμε επίσης και την Ταϊουάν. Η Ταϊουάν επίσης η κατασκευή που είναι πάρα πολύ σημαντική, ο κατασκευαστικός τομέας για την τεχνολογία 5G. Οι μεγάλες ε, εταιρείες εκεί είναι σημαντικές για την οικονομία α, της τεχνολογίας 5G. Οι υπόλοιπε χώρες του κόσμου θα είναι κυρίως καταναλωτές. Ποιοι είναι λοιπόν οι κινητήριοι μοχλοί για αυτή την πολιτικο-οικονομική θέση. Αποτελούνται από τρία στοιχεία. Από τη μία έχουμε τις πιέσεις της βιομηχανίας των προμηθευτών. Και έχουμε και την αποδοχή των ε, φορέων κινητής τηλεφωνίας. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία οι φορεί παροχής κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν και πολλές επιλογές. Είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ασία γίνεται παραγωγή του... Υπάρχει το ακόλουθο μοντέλο. Η κυβέρνηση έχει τη βιομηχανική πολιτική η οποία οθεί και τους προμηθευτές. Στην Κορέα είδαμε ακριβώς αυτήν την καινοτομία να λαμβάνει χώρο όταν είχαμε το, το upgrade από το 3G στο 4G. Είναι, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς έλαβε χώρα. Στην Κορέα αυτό που κάνουν είναι να δίνουν πολύ μεγάλη φορολογική στήριξη, φορολογικές διευκολύνσεις. Το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών οθείται από τους φορείς και από τους προμηθευτές που αυτοί ασκούν πιέσει στην κυβέρνηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τόσο τους προμηθευτές όσο και τους φορείς που ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. Είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο κίνημα marketing αυτή τη στιγμή στην ε, Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αυτή είναι μια παγκόσμια τεχνολογία που είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και διακυβεύονται βεβαίως τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό που λέμε δει μεχρι στιγμης και διακυβευονται βεβαίω τεραστια είναι Αφενός υπάρχει βραχυπρόθεσμη οπτική γωνία, όπου η τεχνολογία 5G θα είναι συμπληρωματική άλλων γενεών κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi, σε μικρά δίκτυα, σε αστικά τοπία σε, με τεράστιο κόστος. Η μακροπρόθεσμη οπτική που θα πρέπει θεωρώ να ακολουθήσουμε είναι ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή 5G σε πάρα μα πάρα πολλού τομεί. Δεν έχουμε χρόνο να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες και παραδείγματα τώρα, αλλά παρόλα αυτά η τεχνολογία αυτή 5G θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ιδού λοιπόν και τα συμπεράσματά μας. Τι έχουμε στα χέρια μας. Τα επιχειρηματικά μοντέλα δεν είναι σαφή. Αυτό είναι το, το πρώτο συμπέρασμα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, η ζήτηση στην αγορά επίσης είναι αβέβαιη. Οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από ό,τι για τις προηγούμενες γενιές α, τεχνολογίας Άρα δεν είναι σαφές ποιος θα επενδύσει και ποιος θα πληρώσει το κόστος. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή ο θόρυβος γύρω από την τεχνολογία είναι τεράστιος. Πρόκειται για μια περίπτωση ρούχων του αυτοκράτορα. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Η ο ενθουσιασμός από τους ήδη υπάρχοντες πάροχους κινητή τηλεφωνίας μπορεί και να έχει υπερεκτιμηθεί. Ποιες είναι οι συστάσεις μας. Μακροπρόθεσμη τεχνολογική έρευνα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξαπλωθεί η τεχνολογία αυτή. Θα πρέπει να γίνουν λεπτομερείς μελέτες των επιχειρηματικών μοντέλων. Είναι πραγματικά απαραίτητο. Το θέμα με τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι ότι το κόστος είναι τεράστιο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος αυτό. Δεν είναι εύκολο με δεδομένη την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας αυτής. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική για τα δίκτυα 5G που να βασίζεται στην ενθάρρυνση της κοινή χρήση υποδομής και στον διαχωρισμό υποδομής και υπηρεσιών. Το βλέπουμε μέχρι σε ενό σημείου στη Σιγκαπούρη αυτό, αλλά και στην Κίνα, όπου ένα συγκεκριμένο δικτυο δίκτυο 5G μπορεί να μειώσει το κόστος των φορέων παροχής κινητής τηλεφωνίας. Αυτό που ελπίζουμε, αυτό που ευελπιστούμε ότι θα συμβεί, είναι να συντονιστούν οι προσπάθειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να ξεκινήσουμε με περιορισμένη ε, κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Ε, έχουμε μία μικρή καθυστέρηση και θα πρέπει να περιορίσω το χρόνο Και να ξεκινήσω με τους συντονιστές, ε, εκπροσώπους των συντονιστών έστω. Η κυρία Καρβάλιο. Δύο λεπτά έχετε ο καθένας. Κυρία Καρβάλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση να τονίσουμε τη σημασία του 5G, να τονίσουμε τη σημασία για την Ευρώπη, για τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ανταγωνιστικότητά της, γιατί θέλουμε να είμαστε ηγετικοί Ήπριος στην τεχνολογία αυτή. Δύο ερωτήσει. Είπατε στην ερευνά σας ότι είναι κλειδί το μέγεθος και η κλίμακα της συνολικής αγοράς. Στην παρούσα φάση, όπου δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η τυποποίηση, θα είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία ισχυρή ευρωπαϊκή εγχώρια αγορά, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το αναφέρεται μεν στην έκθεση, αλλά δεν βασική σας σύσταση στα τελικά σας σχόλια. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με την πρώτη. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις ε, ΗΠΑ και με την Κίνα. Ξέρουμε ότι διάφορα κράτη-μέλη της Κίνας ε, έχουν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Κίνα, κυρίως. Πώς πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει την ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αγοράς. Μήπως αυτό προκαλέσει πιο μεγάλο κατακαιρματισμό. Και ποια θα πρέπει να είναι η προσέγγισή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αυτές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Είπατε στην αρχή της παρουσίασής σας ότι υπάρχει έλλειψη τυποποίησης ενός ομογενούς χαρακτήρα. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε μία τέτοια τεχνολογία, δίκτυα πολλών δισεκατομμυρίων, χωρίς να ξέρουμε τις προτεγραφές που χρειάζεται να τηρούμε. Γιατί πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εκχώρησης τέτοιων συμβάσεων. Αλλά με τι προδιαγραφές. Δεν υπάρχει λοιπόν η σχετική τεχνολογική οριμότητα. Δεν ξέρουν τι δίκτυο χρειάζεται. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην ε, Επιτροπή αυτή στην προηγούμενη θητεία προσπαθήσαμε να αποφύγουμε πολύ τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί κατά την ανάπτυξη του δικτύου 4G. Και είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε τεχνικέ υπερογραφέ, να υπάρχει οργάνωση στα κρατημέλη κτλ. Έχετε πει δύο λόγια για το πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε τώρα όμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση και μία τρίτη ερώτηση. Πιστεύετε αυτή η έλλειψη όρεξης, αν θέλετε, για την ανάπτυξη του δικτύου 5G από πλευρά των επιχειρήσεων. Γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πού θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Αλλά η έλλειψη εφαρμογών, χρήσης 5G. Πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. σε ό,τι αφορά και την έλλειψη χρηματοδότησης. Και ε, τέταρτη ερώτηση για την Huawei. Θα πρέπει να υπαχθεί σε ξεχωριστή ε, ρύθμιση. Είναι σημαντικό θεωρώ το ερώτημα αυτό στην Επιτροπή Ήτρε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, η κυρία Κλαμπάιωβα. Ο συνάδελφος θα κάνει την ερώτηση ο κύριος ε, Φλέγκο. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Ελπίζω όλοι να ωφεληθήκατε όσο και εγώ από την παρουσίαση αυτή. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο του μιλητή. Συνεχίζει τώρα. Είχα λοιπόν την τιμή να παρευρεθώ στην Κίνα και να επισκεφθώ ε, τα κεντρικά της Huawei και είδαμε πόσο προωθεί η κινέζικη κυβέρνηση την εταιρεία αυτή στον τομέα της ε, καινοτομία και τη ανάπτυξη, τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε κορυφαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοια ζητήματα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επενδύουμε πιο πολύ στην έρευνα. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω το εξή, να κάνω μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το 5G, σε ό,τι αφορά τους σταθμούς ε, και τους κεραίε, κεραίες, τους Τα πράγματα είναι πάντα περίπλοκα. Υπάρχουν λοιπόν πρότυπα σε σχέση με την τρέχουσα τεχνολογία σε ό,τι αφορά και τους ε, σταθμούς ή μήπω ακούμε πιο πολύ ζητήματα marketing ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μπούχνερ. Από τους πράσινους, ο κύριος Μπούχνερ. να αναφέρω καταρχάς το εξής. Τα εμπορικά συμφέροντα ε, πάντα είναι, παίζουν ένα ε, ρόλο. Να σας αναφέρω τον κύριο Μπάνι, ο οποίος στο Γερμανικό Κοινοβούλιο είπε στις 3 Ιουλίου ότι θέλετε να έχετε πληροφορίες για τα πάντα. Μιλάμε για πολιταρχικές τέτοιες ε, αντιμετωπίσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την συγκέντρωση στοιχείων για θέματα τρομοκρατία. Ουσιαστικά συγκεντρώνουμε ε, στοιχεία για τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους που μένουν στον πλανήτη μας. Αυτό λοιπόν γίνεται μόνο με το 5G. Μιλάμε λοιπόν για τεράστια εμπορικά συμφέροντα, αποκλειστικά εμπορικά συμφέροντα. Να μην ε, ξεχνάμε ότι αυτά θα επικρατήσουν σε ό,τι αφορά τους χρήστες και έχουμε και πολιτικά, ε, πολιτικές επιρροές ό,τι αφορά τα εμπορικά συμφέροντα. Αυτό που επίσης ε, αποτελεί παράγοντα είναι το θέμα της υγείας και το κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε τουλάχιστον δύο μηχανισμούς πρόκλησης βλαβών στην υγεία από την τεχνολογία 5G. Αυτό δεν αναφέρθηκε λοιπόν και έλειψε από την παρουσίαση και θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Και τέλος, από την έκθεση μου λείπουν και οι εναλλακτικέ που υπάρχουν αν θέλουμε να μεταβούμε σε πιο υψηλές συχνότητες. Thank you Ευχαριστώ, Μπόρκια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για τους δύο καθηγητές για την εξαιρετική σας ε, παρουσίαση. Ο οι συνάδελφοι Μπούχνα και Φλεώση εν μέρη κάλυψαν ε, τη δική μου ερώτηση. Είναι αναμφίβολο ότι σε επίπεδο κοινή γνώμη ε, επικρατούν μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία από την ανάπτυξη των δικτύων Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή αν έχει υπάρξει κάποια ε, λύση ή αν υπάρχουν σχέδια μελέτηση για αυτά τα θέματα. Έχουν μάλιστα ε, υποβληθεί σχετικές ερωτήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά το θέμα της ψηφιακής εξάρτησης, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την παιδική ηλικία και γενικά τους ε, νεότερους. Η μελέτη θα αναλύσει και το θέμα της ψηφιακής εξάρτησης ε, και όλος ιδιαίτερος όσον αφορά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ξανθαντάσκη. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Η μία αναφέρθηκε ήδη. Το γεγονό ότι τα δίκτυα 5G θα είναι πολύ πιο πυκνά σε σχέση με τα υφιστάμενα δίκτυα και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα έχουν επιρροή σε ό,τι αφορά τα πρότυπα για την γραμματική ακτινοβολία. Και στη χώρα μου κυρίως υπάρχουν μεγάλες, ε, μεγάλη δισταγμή. Τι και το θέμα της ε, κοινωνικής αποδοχής του δικτύου 5G. Αυτό αφενός. Δεύτερη ερώτηση, το θέμα της ε, ασφάλειας δεν έχει αναφερθεί καθόλου. Η κυβέρνηση μου έχει προσυπογράψει μια σχετική διακήρυξη, δήλωση με τις ΕΠΑ. Και ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα του κατά πόσον μπορεί να υπάρξει καν ασφάλεια επαρκής σε δικτυα 5G. Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα δηλαδή. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δισταγμοί και αμφιβολίες σε ό,τι αφορά και τη δραστηριοποίηση κινέζικων επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Γιατί θα κλείσει ο κατάλογος. Ναι, ναι, και εσείς, και εσείς. Ένα λεπτό έκαστος. Κυρία Δερκαστήγιο. Ευχαριστώ. Εξαιρετική έκταση. Και χρειαζόμαστε τέτοιες ε, έρευνες. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση περίπλοκη. Ένα βήμα, δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω. Πάντα ανακύπτουν προβλήματα. διαρκώς, πέρα από τα προβλήματα, τα ιατρικά. Έχουμε κάνει διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά την υποδομή. Πολλά έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά την υποδομή. Το ECC, e κώδικα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, υπάρχουν προδιαγραφέ για τέτοιες χρήσεις για την πώληση των ε, κινητών τηλεφώνων και το καταξής. Αν λοιπόν μπορούσατε πέρα από όλα αυτά να προτείνετε δύο-τρία μέτρα τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλό θα ήταν να αποφασιστούν. Βράχει πρόθεσμα, άμεσα. Ποια θα ήταν τα μέτρα αυτά. Πιο πολύ σε σχέση με την έρευνα, τη χρηματοδότηση, τις υποδομές. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπετε, και χρειάζεται να υιοθετήσουμε τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ. Κύριε Κομπουλάντρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ήταν και πιο σκεπτικιστική σε σχέση με άλλες τέτοιες παρουσιάσεις. Οι συστάσεις ήταν όμως λίγο πολύ ίδιες με άλλες. Πείτε μας λοιπόν γιατί ήσασταν τόσο διστακτικοί και παρόλα αυτά στις συστάσεις λέτε εντάξει, πράσινο φως. Να συνεχίσουμε. Αν σωστά κατάλαβα τουλάχιστον αυτό είπατε. Τα τελευταία πέντε έτη που συμμετείχα και στην ε, χάραξη της νομοθεσίας είδαμε ότι το 4G ήταν πιο γρήγορο από ότι την τεχνολογική προσαρμογή και το θέμα είναι ότι είμαστε ένα έθνος χρηστών και τελικά το περιεχόμενο μεταφέρεται αλλού, όλα μεταφέρονται αλλού. Και τελικά το θέμα είναι ότι δεν είμαστε εκεί που χρειάζεται. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα της ψηφιακής οικονομίας, γιατί εδώ πέρα μιλάμε μόνο για ψηφιακή υποδομή. Χρειάζεται προφανώς, αν μείνει πίσω η Ευρώπη, τα κοινοτομία, τα οικοσυστήματα θα μεταφορθούν αλλού. Και εμείς θα καταλήξουμε να είμαστε ένα έθνος, έθνος χρηστών και μόνο. Αυτό είναι το βασικό μου θέμα και το τονίζω ότι η λογική συνέπεια στα τέρα θα πρέπει να επενδύουμε διαρκώς στα δίκτυα αυτά προκειμένου να προχωρήσουμε αυτόματα στο 5G γιατί μόλις σταματήσουν οι επενδύσεις θα μείνουμε πίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος είναι. Ένα λεπτό έχει στη διάθεσή σας. Θα μιλήσω στα φιλανδικά, τη γλώσσα μου, αν μου επιτρέπετε. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και ε, καταλαβαίνω ότι το 5G στην πράξη σημαίνει ότι το σήμα από τους σταθμούς θα πρέπει να κινείται σε λιγότερες, μικρότερες αποστάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες. Στην Ευρώπη έχουμε αρακοτακημένες περιοχές. Αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση αν θέλουμε να καλύψουμε πραγματικά το σύνολο της Ευρώπης. Τι είδους προκλήσεις λοιπόν διακρίνεται στο σημείο αυτό. Όταν θα θελήσουμε να εφαρμόσουμε το 5G θα πρέπει να γίνουν λοιπόν τεράστιες επενδύσεις σε, σε δίκτυα, σε σταθμούς. Πέρα από αυτό πιστεύετε ότι υπάρχουν προβλήματα άλλα. Ευχαριστώ. Η κυρία Παύλους, τελευταία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. και την έρευνά σας. Ένα σημαντικό στοιχείο μου λείπει. Το θέμα της βιωσιμότητας. Αν λάβουμε υπόψη ότι απότερο στόχος μας θα πρέπει να είναι ε, η μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς την εκπομπή άνθρακα. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε γρήγορα. Υπάρχουν λοιπόν ε, οποιαδήποτε εκτιμήσεις ε, αν υπήρχε πραγματικά μεγάλες κλίμακες ανάπτυξη της, ε, του 5G, του 5G. Και αυτό πώς θα ενταχθεί στο στόχο για την κλιματική ουδετερότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει το λόγο. Ο κύριος Μπλάκμαν, να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε για την έρευνά μας. Να σας ευχαριστήσω και για τις ερωτήσεις σας που καλύπτουν ε, μεγάλο φάσμα θεμάτων. Να προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες εξ αυτών και ο Σάιμον στη συνέχεια μπορεί να πάρει το λόγο να απαντήσει τις υπόλοιπε. Δεν τις ε, απαντάω με την σειρά της ερωτήσεις, αλλά ουσιαστικά το αναπάντητο ερώτημα που παραμένει είναι Ποιος είναι ο σκοπός του 5G, γιατί χρειάζεται. Άρα πολλά έχουν να κάνουν με αυτό. Η ίδια μηχανία ψάχνει φυσικά νέες ε, πηγές προσόδων και προφανώς τα σπρώχνει όλα αυτά. Αλλά δεν είναι σαφές για το τι προορίζεται αυτή η τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη αυτή η τεχνολογία σε σχέση με την προηγούμενη. Έχουν πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και γίνονται διάφορες ε, δοκιμές, πειράματα. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το τρέξουμε γρήγορα και βιαστικά. Να έχετε υπόψη σας αυτά που λέγαμε και να είσαστε και λίγο διστακτικοί για αυτά που προωθούνται. Θα υπάρχουν ε, μεγάλα ωφέλη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα ωφέλη αυτά, αλλά Βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασίας. Όταν βλέπουμε λοιπόν διάφορους ε, ε, φορεί εκμετάλλευση εκμετάλλευσης που προωθούν διάφορα στοιχεία, διάφορες εφαρμογές για το 5G, ουσιαστικά δεν είναι 5G αυτά που προωθούν, είναι 4G, άντε 4,5G το πολύ. Άρα δεν χρειάζεται να βιαστούμε, αυτό λέμε. Χρειάζεται να κάνουμε έρευνα, να σκεφτούμε καλά της χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Όχι απλά να πετάξουμε χρήματα σε ένα κουβά και τελικά να μην ξέρουμε ποια θα είναι τα πλονεκτήματα και τα ωφέλη. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. Άρα είμαστε διστακτικοί. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να το βάλουμε κατά μέρο. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει όμως μια μακροπρόθεσμη ε, νοοτροπία και να τα σκεφτούμε καλά όλα αυτά. Αναφέρατε πολλοί από εσάς θέματα υγείας και ενδεχόμενο ρίσκο κίνδυνο για την υγεία. Σε μια σύντομη τέτοια έκθεση αναφέρουμε κάποια στοιχεία για την υγεία. Αν και προφανώς είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι ο Σάιμον θα τα απαντήσει καλύτερα αυτά για το θέμα της υγείας δηλαδή. γιατί το εξετάζουμε αυτό σε σχέση και με ένα άλλο project το οποίο προετοιμάζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για τον, την ανάπτυξη μικροδικτύων. Τι άλλο να σας πω. Σάιμον, θες να πάρεις το λόγο να απαντήσεις και εσύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις που έγιναν για τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές συγκείμενο, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας ε, μεγάλης τεχνολογίας, πολύ σημαντικής τεχνολογίας για όλο τον κόσμο. Και όταν μου είδα τα σχέδια για την τεχνολογία 5G, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι δεν θα ξεκινήσω από εκεί, αν θα ήθελα να πετύχω το σκοπό αυτό. Και όσοι εφαρμόζουν την 5G, τεχνολογία 5G, και πάλι δεν χρησιμοποιούν τόσο υψηλές συχνότητες, χρησιμοποιούν αυτό το μεσαίο φάσμα, το μέτριο φάσμα, γύρω στο 1 GHz. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά χρειάζονται πολύ λιγότεροι σταθμοί. Όταν κοιτάμε λοιπόν υψηλέ συχνότητε για πυκνοκατοικημένε αστικές περιοχές, ουσιαστικά για αυτούς έχει σχεδιαστεί το σύστημα. Άρα το ερώτημα της Φιλανδίας ήταν πολύ εύστοχο. Μιλάμε λοιπόν για μια τεχνολογία η οποία κάπως είναι μονόπλευρη Χρειαζόμαστε πιο πολύ έρευνα και ανάπτυξη, γιατί αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε φάσματα πολλαπλών συχνοτήτων για να έχουμε ε, καλύτερη κάλυψη για αριακοτοικημένε περιοχέ σε χαμηλό κόστο, θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτό με οδηγεί με τη σειρά του στα προβλήματα υγεία, τα οποία ενδεχομένω να προκληθούν. Γιατί τα πεδία διάδοση που βλέπουμε σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία 5G είναι πολύ διαφορετικά από τις τροπικές ε, κεραίες που χρησιμοποιούμε ως τώρα, που είναι μονοπλευρές. Χρειαζόμαστε λοιπόν, ε, ως τώρα μάλλον σήμερα, όχι μόνο το χρόνο και την ε, συχνότητα, αλλά και τον χώρο. Και έχουμε λοιπόν κτίνες οι οποίες ε, ε, για να κινηθούν με τέτοια ταχύτητα και να είναι και κατανοητές και ευδιάκριτες, θα πρέπει να είναι πολύ πιο πυκνές. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε προβλήματα για την υγεία. Όσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα λοιπόν, η διείσδυση στον ανθρώπινο ιστό μικραίνει. Άρα είναι πιο ασφαλές το δίκτυο αυτό το ακούμε συχνά και κάτι άλλο που ακούμε είναι ότι αν υπάρχει πυκνή κάλυψη και ανάπτυξη θα έχουμε δύο πεδία, το πεδίο των σταθμών αλλά θα έχουμε και τα πεδία από τη συσκευή, την κάθε συσκευή του καθενός. Και η πυκνή λοιπόν ανάπτυξη σε μικρές αποστάσεις θα μειωθεί και αυτό θα επηρεάσει το άνατο πεδίο το οποίο μπορεί κανείς ε, να δεχτεί. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του 5G. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό και γι' αυτό λοιπόν αναφέρουμε και τον σκεπτικισμό. Είμαστε προσεκτικοί και αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι χρειάζεται πολύ παραπάνω δουλειά. Πρέπει να εργαστούμε πολύ πιο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι την τεχνολογία αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε πιο πολύ στα εργαστήρια και μετά επιτόπου. Χρειαζόμαστε μέτρηση επιτόπου, όχι ε, μέτρηση σε διάφορα εργαστήρια για την, ε, ε διάδοση και την εξάπλωση. Και αυτό με οδηγεί λοιπόν με ωραίο τρόπο στην ερώτηση του ποιος ε, τελικά κερδίζει και ποιος χάνει σε αυτή την, αυτόν τον αγώνα του 5G. Αυτό το έθεσαν πολύ ω ερώτημα και ποιε είναι και οι σχέσει μα με τον υπόλοιπο κόσμο, μήπω προκαλείται καταγραμματισμό. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Αν κοιτάξουμε διάφορε ευρεσιτεχνίε οι οποίε έχουν ε, χορηγηθεί, η Ευρώπη τι χρειάζεται καταρχά. Α, μάλλον η Ευρώπη έχει την Νόκια στο πρώτο θέμα. Αλλά στι εφαρμοσμένε ε, ευρεσιτεχνίε είναι Huawei πρώτη, γιατί είναι τεράστια σε ό,τι αφορά τι ευρεσιτεχνίε έχουν ζητήσει πάνω από χίλιε και έχουν ε, πάρει μόνο 74 ευρεσιτεχνίε. Άρα εδώ πέρα υπάρχει με διάφορα σε σχέση με τις ε, ευρεσιτεχνίε που έχουν ζητηθεί και έχουν χορηγηθεί. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα στι εμπορικέ στις εμπορικές τεχνολογίες. Τι κάνουμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και αγοράζουν ε, πατέντε και μετά τα βάζουν σε πακέτα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι κάποιε βασικέ ευρεσιτεχνίε, οι οποίε είναι απαραίτητε για την ανάπτυξη δικτύων 5G. Το θέμα λοιπόν είναι να ελέγξουν ακριβώ αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και προφανώ είναι τεράστιε οι νομικέ διαμάχε που γίνονται και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια θέματα, για τη χρήση ακριβώ των ευρεσιτεχνιών αυτών και κατά πόσον είναι πραγματικά σωστή η χρήση τους και δικαιολογημένη. Και αυτές τις μάχες τις βλέπουμε για παράδειγμα και στην Apple. Όταν λοιπόν περνάμε σε θέματα 5G, ουσιαστικά πρόκειται για μία μάχη των ευρεσιτεχνιών. Όταν κοιτάξουμε λοιπόν τελικά ποιο θα ωφεληθεί και ποιο θα χάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν χάνουμε. Η Ericsson είναι στην πέμπτη έκτη θέση σε ό,τι αφορά τι πατέντε, κάπου στο μεταξύ είναι και οι Αμερικάνοι η Samsung είναι μεταξύ των πρώτων και οι Κορεάτες θα πάνε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της καινοτομίας μέσω των ευρωστεχνιών. Άρα δεν θεωρούμε ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε καμία περίπτωση. Για μία άλλη ερώτηση. Το θέμα το οποίο κανείς δεν θέλει να αναφέρει ποια θα πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με την Αμερική και την Κίνα. Η Huawei παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Το συζητήσαμε λοιπόν αυτό με τους συναδέλφους και η αρχική μου αντίδραση την οποία την απέρριψε στην απέραντη σοφία του Κόλλιν ε, ε, πάρα αυτά, ήταν ότι δεν έπρεπε να κάνω κανένα σχόλιο εδώ μπροστά σας, αλλά θα κάνω σχόλιο. Αυτό που δεν βλέπετε είναι... Αυτό που μάλλον που βλέπετε δεν είναι η επιχείρηση, είναι η κυβέρνηση πίσω από την επιχείρηση. Αυτό ισχύει και για τους Αμερικάνους και για τους Κινέζους. Είναι πολύ σημαντικό πολιτικό σημείο αυτό τώρα. Ποια κυβέρνηση πιστεύεστε, αν δεν τις εμπιστεύεστε, να ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή τεχνολογία. Γιατί θα πρέπει να εμπιστευτούμε αυτές τις κυβερνήσεις πιο πολύ. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνουν στη χώρα μου σήμερα και αύριο θα είναι πολύ σημαντικά για αυτό που συζητάμε. Γιατί έχουμε πολλά να δώσουμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα δώσουμε, αλλά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να τα δώσουμε. Πρέπει λοιπόν να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζουμε κάπως να κινηθούμε σε σωστά πλαίσια. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε μείνει πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποιους τομείς ηγούμαστε μάλιστα, αλλά σίγουρα δεν έχουμε μείνει πίσω. Θα πρέπει να χρειαστεί ε, μα, κάποια προσαρμογή, αλλά δεν έχουμε μείνει πίσω. Και ζητώ συγγνώμη αν δεν έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμμετοχή σας και για τις ε, παρουσιάσεις σας. Συνάδελφοι, μπορείτε να βρείτε την έκθεση καθώς και την μελέτη. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας. Ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Γενικό Διευθυντή Πακέ σχετικά με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Πακέ Okay, let's start Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Όπως είπα, το επόμενό μας θέμα προσυζήτηση ε, με τον Γενικό Διευθυντή ε, Ρίκ Πλακέ σχετικά με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ Γενικέ που ήρθατε για να συζητήσουμε αυτή τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Είχαμε στην Επιτροπή μας εκθέσεις από τον κύριο Χέλλερ και τον κύριο Νίκα. Βεβαίω για μας το Horizon Europe είναι ένα από τα πιο σημαντικά ε, προγράμματα και μας ενδιαφέρουν πάντοτε και έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για αυτά τα προγράμματα στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την κλίμακα, την ταχύτητα, τον προπολογισμό και γι' αυτό το λόγο Έχουμε φτάσει σε μερική συμφωνία για το Horizon Ευρώπη πριν από τη διακοπή για τις εκλογές και αυτό σημαίνει εκτεταμένες ανταλλαγές απόψεων με το Ευρωκοινοβούλιο για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. <coughs> Γι' αυτό το λόγο και τόσο γρήγορα σας καλέσαμε εδώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ανταποκριθήκατε τόσο γρήγορα. Θα σας δώσω λοιπόν τον λόγο να παρουσιάσετε τις πιο πρόσφατες ενέργειες της Επιτροπής από τότε που διακόψαμε για τις εκλογές και βεβαίως μετά στη συνέχεια οι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να σας υποβάλουν ερωτήσεις και διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχάς έχετε εσείς το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου και προνόμιό μου να απευθύνομαι στην Επιτροπή Ήτρε και βεβαίως ε, εξ ονόματος του ε, Επιτρόπου που θα ήθελε πολύ να είναι σήμερα παρόν, το κύριο Μοέδος. Ε, βεβαίως θα πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αξιοσημείωτη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών που επέτρεψε την πρώιμη πολιτική συμφωνία για το θέμα με τη συνεργασία του Κρίστιαν Έλλαρ και του κ. Νίκα ε, καθώς και τη στήριξη πολλών εξημών στην Επιτροπή. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό γιατί αναμέναμε πολλά, αναμένει πολλά η επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ήταν πολύ σημαντικό για την προετοιμασία του Horizon Ευρώπη, που είναι και το σημερινό μας θέμα σήμερα, θα απαιτήσει διαφόρων ειδών, μάλλον διαφορετικού είδους προετοιμασία από ότι το προηγούμενο πρόγραμμα Horizon 2020. Και το να εκπροετοιμαστούμε έτσι έγκαιρα μας δίνει χρόνο ε, ε, άπλετο για να προετοιμαστούμε για την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο ε, είναι πολύ σημαντικό. Πρόγραμμα που ελπίζουμε πως ε, θα συνοδευτεί από έναν φιλόδοξο ε, προϋπολογισμό βεβαίως και ξέρω πως το και Ευρωκοινοβούλιο είναι ακόμα πιο φιλόδοξο από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα καλύψουμε το ίδιο το πρόγραμμα αν και γνωρίζω πως το κείμενο είναι καινούριο για πολλούς από εσά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα και βεβαίως και θα ε, μας ε, ευχαριστεί το ενδιαφέρον των μελών να κάνουμε συγκεκριμένη συζήτηση. Ίσως θα μπορούσαμε, Ντανίκα και το Κριστιαν, να το διοργανώσουμε αυτό, γιατί το νομικό κείμενο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και κάποιες φορές ε, περίπλοκο, ε, αλλά ελπίζω πως στη συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό θα μπορέσετε να αντιληφθείτε ακριβώς πώς προχωράει ε, το πρόγραμμα και πώς ε, συμφωνείτε με βάση την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον περασμένο Απρίλιο. Έκτοτε λοιπόν έχουμε ενεργά ξεκινήσει την προετοιμασία του Horizon Ευρώπη και ιδιαίτερα είμαστε, δραστηριοποιηθήκαμε για τη σύνταξη ενός στρατηγικού ε, πλάνου που είναι ένα νέο βήμα στο ορίζον ε, Ευρώπη ενδιάμεσα ας πούμε ανάμεσα σε μια νομική πρόταση και την νομική, το νομικό οικοδόμα αλλά και, και το πρόγραμμα εργασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Horizon 2020, εκεί δεν περιλαμβάνεται στρατηγικό σχεδιασμός, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά ε, περίπλοκο ήδη και γι' αυτό τότε ε, προχωρήσαμε άμεσα από το νομικό σχέδιο στο στις προτάσεις που υπευλήθησαν για χρηματοδότηση. Η επιλογή τώρα του συνομοθέτη στο Horizon ε, Ευρώπη. Είναι πιο ανοιχτό κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει τη φιλοδοξία ώστε να γίνει έρευνα και καινοτομία με λιγότερο κατακαιρματισμένο τρόπο, πιο οριζόντιο τρόπο. Γι' αυτό και το νομικό κείμενο είναι πιο ευέλικτο και άρα απαιτεί επιπλέον δουλειά. Και Βεβαίω γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η φάση του στρατηγικού σχεδιασμού. Και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν για την στενή ανάμειξη του Κοινοβουλίου και συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό του στρατηγικού ε, αυτού ε, σχεδίου. Το πρώτο σχέδιο λοιπόν διατέθη για δημόσια διαβούλευση πριν το καλοκαίρι. βεβαίως και στην γραμματεία Ήτρε και είμαι βέβαιος πως θα είχατε την ευκαιρία να το εξετάσετε. Η διαβούλευση συνεχίζεται μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στα τέλη του ε, Σεπτεμβρίου 25 με 26 και 26 Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε ημερίδες ε, καινοτομίας και, ανα, και έρευνας. Σε αυτές ε, συμμετέχετε κι εσείς και είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σας, όπου θα συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο το στρατηγικό σχέδιο θα συζητηθεί με τα κρατη με το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά βεβαίως χρειάζεται να συζητηθεί και με λεπτομέρειες με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ένωση. Οι μέρες ε, έρευνας και κοινοτομίας σχεδιάζονται ακριβώς έτσι ώστε να μπορέσουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής που εργάζονται σε αυτόν τον ε, στρατηγικό σχεδιασμό και οι εθνικοί εκπρόσωποι να έρθουν σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους ε, για το ορίζον 2000, ε, συγγνώμη, ορίζον ε, Ευρώπη, ώστε να υπάρξει στην ουσία συνσχεδιασμός των προτεραιοτήτων εφαρμογής του ορίζον Ευρώπη. Βέβαια, σε συνεργασία με τους δύο συνομοθέτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό θα γίνει λοιπόν στη διάρκεια αυτών των ημερίδων μελέτης για την καινοτομία και την έρευνα παραδοσιακά είχαμε ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, από στις ομάδες εργασίας. Εδώ ε, όμως αποφασίσαμε ότι θα ανοίγαμε τη συνεργασία σε όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων και είχαμε και πάλι εξαιρετικά μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντες όπου χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε σωστά το στρατηγικό σχέδιο που θα καλύπτει το πρώτο, την πρώτη φάση, τρία με τέσσερα χρόνια. Θα ενημερώνεται καθώς θα εφαρμοστεί το ορίζον Ευρώπη και δεν θα στοχεύει στην ε, πλήρη ανάλυση όλων των λεπτομεριών, αλλά θα έχει στόχο τη σύνδεση των προτεραιοτήτων του προγράμματος με τις ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας και ε, καινοτομίας. Και ε, έτσι θα εστιάσει περισσότερο στον αντίκτυπο και όχι στο λεπτομερή ε, οδικό χάρτη, γιατί θέλουμε να αφήσουμε ευελιξία στους ερευνητές μας, στις μικρομεσαίες, ε, να μας πούνε τι καινοτομίες, τι λύσεις μπορούν να προτείνουν ε, με βάση τις προτεραιότητες που θα, έχει θεσπίσει, θα έχουν θεσπίσει οι συνομοθέτες μέσω αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Μετά από τις ημερίδες έρευνας και καινοτομίας θα ενημερώσουμε το έγγραφο και στη συνέχεια, στη διάρκεια του 2020, θα ε, ε, ε, οριστικοποιηθεί υπό τη μορφή εφαρμοστικών πράξεων, ώστε να υιοθετηθούν και τα προγράμματα εργασίας υπό τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Πέρα από αυτό το γενικό πλαίσιο λοιπόν θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε δύο πολύ σημαντικές νέες διαστάσεις του ορίζουν Ευρώπη. Τις, το ΛΕΣ και το ευθυγνωμισμένο τοπίο της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και τις εταιρικές σχέσεις. Αυτά όλα είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού, περιλαμβάνονται στα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόλοιπη ερευνητική προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι αποστολές και εταιρικέ σχέσεις θα στηρίζουν τους στόχους του προγράμματος. Για τις αποστολές, Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή έχει ορίσει πέντε συμβούλια αποστολής ε, τον Ιούλιο που στηρίζουν τώρα τη διαδικασία εντοπισμού στόχων αυτών των αποστολών. Δηλαδή έχουμε μια αποστολή για τους καθαρούς ωκεανούς και τα υδάτινα συστήματα, έχουμε μια αποστολή για τον καρκίνο, μια αποστολή για τα υγιή, ε, τις υγιείς υγιές και τα τρόφιμα, έχουμε μια αποστολή για τις ε, ουδέτερες ε, πόλεις σε άνθρακα και έχουμε λοιπόν αυτούς τους πέντε τομείς αποστολών που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στο Συμβούλιο το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Είναι μεγάλες καινοτομίε των προγραμμάτων αυτών. Είναι ε, φιλοδοξία του Κάρλος Μοέδας, ώστε να εξασφαλιστεί καταρχάς η ανοιχτή διαδικασία και η συζήτηση για να μπορέσουν οι πολίτες να έρθουν πάλι κοντά στην καινοτομία και την έρευνα. Αυτά τα συμβούλια των αποστολών θα είναι ε, διαθέσιμα για να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και να συζητήσουν με το Ευρωκοινοβούλιο και τα μέλη και έπειτα έτσι να στηριχθούν αυτοί οι πολύ σημαντικοί τομείς, πολύ συγκεκριμένοι στόχοι που απασχολούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολιτική λοιπόν διάσταση είναι αυτή των αποστολών. Δεύτερη διάσταση είναι να ε, συνδεθεί η έρευνα και η καινοτομία, η επιστήμη με τις ε, με, τα αποτελέσματα των δημόσιων πολιτικών. Δηλαδή, η αποστολή δεν είναι το να παράγουμε μόνο επιπλέον επιστήμη, επιστημονική γνώση, αλλά να οργανώσουμε την, επιστημο, την επιστήμη, τις επιστημονικές, ε, τα επιστημονικά πορίσματα και τα πορίσματα ερευνών ε, με την πραγματικότητα, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αν πάρουμε το πράγμα του καρκίνου, να σας πω, ένας καθηγητής στην Ολλανδία όταν το συζητήσαμε μου είπε το εξής ότι δηλαδή οι επιστημονικές μου δημοσιεύσεις ποτέ δεν θεράπευσαν έναν, έστω και έναν ασθενή. Το νοσοκομείο, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι και τα φάρμακα είναι αυτά που θεράπευσαν. Άρα λοιπόν, είτε είναι πρόληψη, είτε είναι θεραπεία, δεν ξέρω τι θα συστήσει η, αποστολή. Σήμερα το πρωί είχα επαφή μαζί τους πρώτη φορά, μόλις πριν έρθω σε εσά Πάντως από την αρχές του επόμενου χρόνου ελπίζω πως θα προκύψουν οι στόχοι για τα συμβούλια αυτών των αποστολών. Θα δουλέψουμε πάνω σε μια υποσημονική ατζέντα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να μεταφραστούν σε πολιτικές, δημόσιες πολιτικές, ώστε το, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται να έρθουμε λοιπόν και πάλι σε επαφή με τους πολίτες αλλά και να εξασφαλίσουμε τον αντίκτυπο αυτών μας των προσπαθειών για τους πολίτες. Ε, αναμένουμε λοιπόν πως οι αποστολές αυτές θα είναι πολύ συναρπαστικές και ότι θα συγκεντρώσουν τους πόρους και των μελών του κλάδου κάθε φορά ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αντίκτυπο και απόδοση. Δεύτερη διάσταση τώρα Επιπλέον είναι βέβαια οι εταιρικέ σχέσεις, πολύ σημαντικές για, τον, για τους συνομοθέτες, γιατί βεβαίως είναι αυτές οι προτάσεις να δημιουργηθούν εταιρικέ σχέσεις και τα άρθρα 1.8.7 ε, και 1.8.5 αναφέρονται σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Εργαζόμαστε επί 12 τέτοιων εταιρικών σχέσεων και περιλαμβάνονται σε ένα παράρτημα του εγγράφου στρατηγικού σχεδιασμού. Έχουμε κάνει αντίκτυπο Έχουμε ε, μάλλον συστήσει μελέτη αντικτύπου και στα site μας γίνονται οι σχετικές επαφές και γι' αυτό και βλέπετε ακριβώς τι γίνεται. Όσοι ήθιστε θα πρέπει να γίνουν, όπως σας είπα, μελέτες αντικτύπου και εδώ ε, θα έχουμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς ώστε να προτιμάσουμε ε, μέσα, τι προτάσεις της Επιτροπής μέσα στο 2020-2021. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα λιγότερο θεσμικού χαρακτήρα και εκεί ε, συνεχίζεται η εργασία. Κύριε Πρόεδρε, για να μην μακρηγορήσω πολύ, θα στραφώ στον τρόπο με τον οποίο ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, με τους ευρωβουλευτές. Ε, αυτό ε, έχει ήδη διατυπωθεί σε δηλώσεις. Υπάρχει ανταλλαγή αποστολών ανάμεσα στον πρόεδρο Μπούζεκ και τον επίτροπο Μοέδας για το πώς θέλει να συνεργαστούμε. Βεβαίως, εργαζόμαστε σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοπαραγωγική διαδικασία και Βεβαίως, ε, ο Επίτροπος και το επιτελείο του θέλουν να συνεργαστούν πολύ στενά με την Επιτροπή Ήτρε και τους βουλευτές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε όσο γίνεται σωστότερα το στατικό σχεδιασμό, τις αποστολές και τις εταιρικέ σχέσεις. Είναι περίπλοκη διαδικασία η οποία διέπει πολλέ τομείς πολιτικής όπου ελπίζουμε η καινοτομία όπως σας είπα και η έρευνα να συνδεθούν με τις δημόσιες πολιτικές και εκεί ε, θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Ευρωκοινοβουλίου. Τα έγγραφα λοιπόν αυτά ε, σας γνωστοποιούνται, όπως γνωστοποιούνται και στα κρατη κατά την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Θα ε, είμαστε διαθέσιμοι να έρθουμε σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, κυρία Πρόεδρε, για να συζητήσουμε για το περιεχόμενο με αρχής γενομένης από σήμερα υπήρχε ένα ομάδα εργασίας ε, του Ευρωκοινοβουλίου που ήταν ε, πολύ ε, καλή στη συνεργασία μαζί μας. Εάν αποφασίσετε λοιπόν να ακολουθήσετε αυτό το τρόπο εργασίας, ευχαριστώ εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας, αλλά και θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους δικούς δικούς σας βοηθούς, καθώς και είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε οποιαδήποτε θέλετε τεχνική φύση ενημερωτική ε, συνεδρίαση από το Σεπτέμβριο. Ήδη συμμετέχετε στις ημερίδε. τέλη Σεπτεμβρίου μάλλον, ήδη ε, ξέρετε για αυτές τις ημερίδες ε, και πολλοί από εσά έχετε ήδη ανταποκριθεί και θα συμμετέχετε. 24 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρη και θα έχουμε διοργανώσει μια δεξίωση ε, από πλευρά του Επιτρόπου Μοέδας ώστε να αρχίσει αυτή η ουσιαστική συνεργασία με το Κοινοβούλιο που είναι απαραίτητη ώστε ο στρατηγικός σχεδιασμός να προχωρήσει σωστά. Δεν ε, κάλυψα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, ούτε το Συμβούλιο καινοτομία. Ε, φυσικά και συμμετέχουν στην προετοιμασία και ε, ξέρω πως θα μου υποβάλλετε πολλές ερωτήσεις και είμαι στη διάθεσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο ομιλία σας, γιατί έχουμε λίγο καθυστερήσει. Πρώτο είναι οι κύριος Νίκα και ο κύριος Έλερ. Αλλά ο κύριος ε, Έλερ θα αντικατασταθεί από την κυρία Καρβάλιο σήμερα. Στη συνέχεια θα έχουμε τους συντονιστές. Ο κύριε Νίκα, εφόσον είστε και συντονιστής, να θέλετε να μιλήσετε λίγο παραπάνω και το ίδιο και για την κυρία Καρβάλια. Και μετά στη συνέχεια οι συντονιστές, οι αντικαταστάτες τους θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Catch the Eye για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Κύριε Νίκα, έχετε έξι ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντή για την παρουσίασή σας. Θέλω να ξεκινήσω να σας ευχαριστήσω πρώτα για όλες τις νύχτες που περάσαμε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές από άλλα και από άλλες πολιτικές ομάδες για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουμε. Ήταν πραγματικά χαρά μας να δουλέψουμε μαζί με την ε, Επιτροπή. Στο τέλος αυτό που είναι σημαντικό είναι το αποτέλεσμα και εμείς ως μέλη των πολιτικών ομάδων του ε, Κοινοβουλίου είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί οι φωνές όλων των εμπλεκόμενων μερών έχουν ε, ακουστεί και το τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό και είναι ένα ιδιαίτερα καλό αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι και όλους τους συναδέλφους μου. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ σήμερα και θα εξακολουθήσουν να εργάζονται μέχρι ότου να τελειώσουμε την έκθεση για το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη, γιατί το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και ξέρουμε πόσο υψηλέ είναι οι προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ. Και προσωπικά έχω συνείδηση το πόσο σκληρά εργαστήκατε το καλοκαίρι. Καταλάβ, καταφέρατε να ολοκληρώσετε πολλά κομμάτια που αφορούν την, ε, το στρατηγικό προγραμματισμό και τις αποστολές. Ε, ελπίζουμε ότι θα έχετε την στήριξη που σας χρειάζεται από τον Επίτροπο αλλά και τον προϋπολογισμό των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει Επίσης, να ολοκληρώσουμε και αυτό το ακαθόδε ζήτημα της ευρωπαϊκής συνεργασίας, έχοντας υπόψη μας το, το Brexit. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί ποτέ το Brexit, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Έχω κάποια ερωτήματα για σας, κύριε Γενικέ. Πώς οργανώνει τη δουλειά της η Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις συνεργασίες και τις αποστολές. Αν μπορούμε να έχουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά τις συνεργασίες. Ένα άλλο ερώτημα. Η Επιτροπή κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συνεργίες, συγκεκριμένες ενέργειες. Και να θυμηθούμε ένα από τα βασικά στοιχεία στη συζήτησή μας ήταν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να οργανώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Και τότε θυμάμαι ότι συζητούσαμε κάποιους από τους ε, πιθανούς α, φορείς που θα μπορούσαν να λάβουν ε, επιδότηση από το πρόγραμμα. Και τότε θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε σεμινάρια, θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε ημερίδες, ούτω ώστε να, να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν αιτήσει, να καταλαβαίνουν τις διαδικασίες, να καταλαβαίνουν τις γρήγορες διαδικασίες, να καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι το IC. Πολλά πολλά σημεία κλειδιά και είχαμε πει τότε ότι δεν συζητάμε για Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και με καθηγητές εδώ πέρα στην Ευρώπη που δεν ξέρανε πώς να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα αυτά από τους τομείς της υγείας, για παράδειγμα, την έρευνα στο τομέα της υγείας. Αυτό που ρωτάω λοιπόν είναι αν σκοπεύετε να κάνετε κάποια έρευνα σε ό,τι αφορά την οργάνωση τέτοιου τύπου συνεδρίων. Πώς εσείς φαντάζεστε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι οι δυνατοί συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αιτήσει για επιδοτήσεις από το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Το τελευταίο μου σχόλιο τώρα. Θυμηθείτε τη διατύπωση που έχουμε στο Horizon Ευρώπη λέμε ότι θα υπάρξει μια εκτενής ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Πώς τη φαντάζεστε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει στην, ε, στις διαδικασίες των εργασιών το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στα πρώτα στάδια του, του προγράμματος. Αυτά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρβάλιο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Πακέ για την παρουσίασή του και για όλη την ε, συνεργασία και συγχαρητήρια όλας για την εξαιρετική εργασία σας αλλά και στον Επίτροπο Μοέμπας. Μπορείτε να βασίζεστε σε μας για να ολοκληρώσουμε με έναν φιλόδοξο και γρήγορο τρόπο όλα αυτά τα οποία ακόμη μας λείπουν. Έχω δύο ερωτήματα εκ μέρους της κυρίας Έλερ, της εισηγήτριας, του κυρίου Έλλερ, του εισηγητή, με συγχωρείτε. Το πρώτο ερώτημα ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Νίκα. Έχει να κάνει με την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου στην ε, νομοθεσία του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη είναι σαφές ότι θα υπάρξει μια εκτενής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όπως αυτή που έχετε με τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ανάλογος τρόπος που θα γίνει αυτή η ανταλλαγή με το Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας αρκετούς τρόπους που θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτές τις ημερίδες έρευνας και καινοτομίας. Αλλά το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και θα θέλαμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση του πώς προβλέπεται να λαμβάνει η χώρα αυτή η ανταλλαγή μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το πιλωτικό σχέδιο, το πιλωτικό ε, το πιλωτικό σχέδιο που ήταν και μέρος των ε, τριμερών ε, διαβουλεύσεων και το στήριξαν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Η ιδέα η βασική ήταν κομμάτι της συμφωνίας. Και ε, συμπεριλήφθηκε και ως τροπολογία που συνυπέγραψαν ο κύριος Έλερ και ο κύριος Νίκα μας έκανε εντύπωση το πώς το αντιμετώπισε η δική σας υπηρεσία. Και είναι σημαντικό για μας το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Γιατί ο κανονισμός βεβαίως είναι κάτι, αλλά η συγκεκριμένη προετοιμασία είναι πολύ σημαντική για να τρέξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Αν μπορούσατε, αν θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό θα μας βοηθούσατε. Ως συντονίστρια τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τρία πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το PDP. Για να έχουμε ένα φιλόδοξο πολιετές δημοσιονομικό πλάνο θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε εσάς είναι τι κάνετε εσείς και Επιτροπή για να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένας τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε φιλόδοξη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία είναι να έχουμε έναν καλό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι, χορηγεί, ότι χρήματα για την καινοτομία βρίσκονται και σε άλλα σημεία του πολιετούς δημοσιονομικού πλάνου. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον κανονισμό συμβατό μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Πώς θα, ποιοι θα είναι λοιπόν οι συγκεκριμένοι ε, όροι για να το καταφέρουμε αυτό. Το δεύτερο ερώτημα επίσης έχει να κάνει με το στρατηγικό σχέδιο, αλλά με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Το γεγονός ότι ζητάμε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο είναι γιατί αυτό είναι ένας τρόπος να συμπεριλάβουμε και ολόκληρη την Ευρώπη. Καλύπτουμε την Ευρώπη, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως η συμμετοχή των πολιτών μας που εξασφαλίζεται μέσω του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις αποστολές, για παράδειγμα, ή τις συνεργασίες, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα όργανα αυτά λειτουργούν με διαφάνεια και ότι δεν θα διευρύνουν το χάσμα που ήδη υπάρχει στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικό, αλλά ακόμη δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρη την έκταση της Ευρώπης. Υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι τρόποι να ορίσουμε τις αποστολές, να ορίσουμε τις συνεργασίες που σε μερικές περιπτώσεις ευνοούν τα εμπλεκόμενα μέρη που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, γιατί κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να έρθουν να συμμετάσχουν στις ημερίδες. Είναι πιο δύσκολο. Είναι καλά αυτά τα όσα έχετε κάνει, αλλά είναι ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να συμμετάσχουμε ως Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα αυτά θα είναι ανοιχτά και θα είναι διαφανή και ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε το χάσμα αυτό αντί να το διευρύνουμε. Και το τελευταίο, το τελευταίο μου σχόλιο έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Έρευνας και το Ινστιτούτο Καινοτομίας. Τι θα γίνει με αυτά τα δύο Ινστιτούτα. Θέλουμε να ενδυναμωθούν τα δύο αυτά Ινστιτούτα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταλαμπάιωβα. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ τον ε, Γενικό Διευθυντή. Σας καλωσορίζουμε αυτή τη Δευτέρα εδώ στην Επιτροπή μας. Σίγουρα παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Ορίζον Ευρώπη ότι ε, η ομάδα η πολιτική ομάδα Μουρινού είναι ιδιαίτερα θερμός υποστηρικτής του προγράμματος. Βεβαίως είναι πάρα πάρα πολύ πολύπλοκο να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε όλα, όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται ε, ως φιλοδοξίες στο, σχέδιο αυτό, στο πρόγραμμα αυτό. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο για σας και για τους συναδέλφους σας, το καταλαβαίνω αυτό που σημαίνει ότι υπάρχει και πολλή δουλειά μπροστά μας. Συνεργίες, προϋπολογισμός, κυρίως οι συνεργίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές συνεργίες με άλλα προγράμματα. Και βεβαίως τη συμμετοχή ε, τρίτων χωρών. Αυτό το τελευταίο ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για, το, για την ομάδα μου, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο και θέλουμε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, τι είδους σενάρια προετοιμάζετε. Ε, και όπως είπε και ο εισηγητής κύριος Νίκα, σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχέδιο και εγώ θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η εκτενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι θα κρατήσετε την υπόσχεσή σας ε, και θα σας ε, βλέπουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σας και τους συναδέλφους σας συχνά. Το τελευταίο σημείο θέλω να ευχηθώ και σε εσά και σε όλους εμάς να μπορέσουμε να βρούμε έναν επίτροπο που να είναι εξίσου ενθουσιάδης όσο ο Κάρλος Μοέντα σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Κάτι το οποίο με φέρνει στο επόμενο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί στο πορτφόλιο του Επιτρόπου. Τι πιστεύετε εσείς, ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος, η κυρία Ντόλντεν. Ευχαριστώ που ήρθατε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας σήμερα. Χαίρομαι ε, που η εφαρμογή του Horizon Ευρώπη επιτέλους έχει δρομολογηθεί και συζητάμε την πρόοδο του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν τεράστια τεράστιες προκλήσεις και η έρευνα και η καινοτομία θα βοηθήσουν. Και βεβαίως αναφέρομαι κυρίως στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε θέματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι το ορίζον Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει την καταπολέμηση των ζητημάτων αυτών, θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, όπως ήδη είπαν και οι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να εφιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη συμπερίληψης του Ευρωκοινοβουλίου στην διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως είπαν οι συνάδελφοι και στην προηγούμενη Επιτροπή και τώρα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, αλλά και στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου. Αν μπορούμε να είμαστε ενημερωμένοι και να συμμετέχουμε, τότε θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι και οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες ε, συμπεριλαμβάνονται στη διαμόρφωση του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Και γι' αυτό το λόγο μέσα από μια πιο συγκεκριμένη ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βοηθήσει. Πώς ακριβώς λοιπόν θα γίνει αυτό, Ένα τακτικός διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Δευτερευόντω, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την ενσωμάτωση ε, του θέματος τη κλιματική αλλαγή, τη διάσταση κλιματική αλλαγή. το πρόγραμμα θα, δεν θα καταφέρει να επιτύχει τον στόχο του 35%. Τι στοχεύει να κάνει η Επιτροπή για να μπορέσουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να επιτύχουμε το στόχο του προϋπολογισμού 35% για το κλίμα. Ο κύριος Πόρκια έχει το λόγο. Ή όποιος τον αντικαθιστά. Ο κύριος Κάζαντέψκι τότε σκιώδης εισηγητής. Έχετε δύο λεπτά. Να μιλήσω τη γλώσσα μου, για να είμαι πιο σαφής. Ως και όταν ε, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε συζητήσεις σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα Ευρώπη. Και πραγματικά δεν είναι καθόλου απλό το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ, ε, πολύ σύνθετο και χάρη στη βοήθεια του συναδέλφων Νίκα και Κέλλερ καταφέσαμε να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά και την αναφορά ε, στις τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής για να ρωτήσω λοιπόν κάτι απλό. Σε τι βαθμό η στρατηγική σας ο στρατηγικός σας σχεδιασμός θα επικεντρωθεί σε τέτοιες ε, περιοχές. Ιδιαίτερα στην οικονομία μετά την ε, ουδετερότητα του άνθρακα και με το ενεργειακό πακέτο θα υπάρξει μεγάλη πίεση η οποία θα γίνει αισθητή σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω λοιπόν ότι η έρευνα και η ανάπτυξη θα πρέπει να παίξουν μεγάλο ρόλο εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εκτιμώ ιδιαίτερω τη συζήτηση η οποία ξεκίνησε για όλο τον ορίζοντα Ευρώπη. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ κυρία Ματίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, εδώ είμαι. Γεια σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ και το επιτελείο σας ε, με τους οποίους ε, διαπραγματευόμαστε αυτά τα προγράμματα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση γιατί συμφωνώ με πολλές άλλες που υπευλήθησαν και έχει να κάνει με το θέμα που μας φέρατε σήμερα, δηλαδή το στρατηγικό σχεδιασμό ε, για το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με μια ανησυχία που ανέκαθεν αναφέρομαι και έχει να κάνει με την εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος του ορίζοντας 2020 είναι το γεγονός ότι είχαμε άνεση συμμετοχή των διαφόρων χωρών όχι μόνο όσον αφορά την κατανομή των πόρων για την ε, καινοτομία και την έρευνα, αλλά και όσον αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχή στην επεξεργασία, στην εκπόνηση των προγραμμάτων και ε, στην εφαρμογή αυτών. Και σε αυτή, από αυτή την άποψη, εφόσον είμαστε ακόμα στη φάση της διαβούλευσης και πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτή η online διαβούλευση ε, με το ευρύ κοινό στις 8 Σεπτεμβρίου, θέλω να σας ρωτήσω τι κάνατε για να καλύψετε στη διάρκεια αυτού της διαδικασίας για να διορθώσετε κάποια από αυτά τα προβλήματα που είχαμε αναφέρει για το Horizon 2020 και για τα προγράμματα πλαίσια, τα αρχαιότερα. Ε, εάν δηλαδή μεριμνήσατε ώστε να υπάρχει μια πιο ισομερής κατανομή ε, συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, ε, πώς το εγγυηθήκατε αυτό και πώς ε, εξελίχθηκε στις διάφορες χώρες γιατί πιστεύουμε πως και αν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να είναι πιο ισότιμο για περισσότερους θεσμούς από περισσότερες χώρες ε, και για να ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά ζητήματα οι πολίτες θα πρέπει από την αρχή, από τη διαβούλευση να υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια ενημέρωση που να ανταποκρίνεται σε αυτό. Ε, ξέρετε λοιπόν τι έγινε ακριβώς, ε, μπορείτε να μας πείτε και έπειτα ποια ήταν η συμμετοχή η δημόσια σε όλη αυτή τη διαδικασία που θα τελειώσει 8 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Και τώρα συνάδελφοι στρέφομαι σε εσά. Ο κύριος Μπούζεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενική Διευθυντά για την ε, παρουσίασή σας. Σας συγχαρητήρια και σε εσά. Ε, να ευχαριστήσουμε και τους ε, συναδέλφους μας, τους συζητητές και τη Ρουμανική Προεδρία, η οποία κατάφερε να ολοκληρώσει τα σημεία αυτά πριν τις εκλογές. Τρία σημεία. Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τεχνολογία και Καινοτομία. Πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του ορίζοντα. Μπορεί να σημαίνει αυτό ενίσχυση αλλά και αποδυνάμωση της υπηρεσίας. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, ε, όπως είπατε, ο ανταγωνισμός θα προωθήσει την ε, καινοτομία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα λάβουμε αυτά υπόψη, γιατί πλέον αυτό είναι στην πλήρη ευθύνη των προγραμμάτων έρευνας και του ε, Επιτρόπου για την έρευνα. Ελπίζουμε λοιπόν να λειτουργήσουν τα πράγματα αυτά πολύ καλύτερα στους κόλπους του ορίζοντα. Δεύτερο θέμα. Είναι σημαντικό από πλευρά ε, της ε, ευρύτερη ε, συμμετοχής, καθότι το EIT ήταν πάρα πολύ δραστηριό στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες. Βοήθησε λοιπόν ιδιαίτερα για να διευρύνει τους ορίζοντες, για να παρακολουθήσουμε Λοιπόν, πώς έγινε αυτή η διαδικασία διεύρυνση, γιατί πετύχαμε μεγάλα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Και τρίτο σημείο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίε του δεύτερου πυλώνα. Θα θέλαμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να συμμετέχουμε σε κάποιες προτάσεις. Γιατί ευρωπαϊκές περιφερειές μας, στις χώρες μας, συναντιόμαστε με τους εκπροσώπους της ε, οικονομίας αυτής. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τους δώσουμε πιο πολλές πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες. Και θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε και πιο πολλές πληροφορίες ε, από ό,τι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις. Πιστεύετε λοιπόν ε, ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο για τέτοιες προτάσεις. Κυρία Τόγια. Για ένα λεπτό. Μάλιστα, ένα λεπτό. Πολύ σύντομα θέλω να θυμίσω επιγραμματικά κάποια θέματα τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι για να σας πω ότι είναι γενικού ε, ενδιαφέροντος. Το είπαν ε, και άλλοι συνάδελφοι διαφόρων ομάδων. Αφορούν το θέμα των σχέσεων με το Κοινοβούλιο. Γιατί και στον εντοπισμό των αποστολών και την ανάπτυξη πιστεύω πως μπορούμε να ε, δώσουμε μια, γενική, μια γενική εικόνα γιατί πρόκειται για αντίκτυπο στον κόσμο. Δηλαδή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα και να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών Έπειτα το θέμα της ε, συνεργασίας υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί πόροι που είναι αφιερωμένοι στην έρευνα και την καινοτομία που ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους ενώ πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τη σύγκληση αλλά και πώς θα, να πούμε στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες πώς πρέπει αυτό να το κάνουμε γιατί διαφορετικά επικρατεί ε, σύγχυση με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες συνεργασίας. Τώρα μιλήσατε για την καινοτομία. Εγώ ανησυχώ ελαφρώς, εν πάση περιπτώσει όχι ακριβώς ανησυχώ, αλλά με προβληματίζει το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα, οικονομικά, τα δημοσιονομικά μέσα. Γιατί ε, είναι σωστό το δημόσιο χρήμα να προσελκύσει το ιδιωτικό χρήμα, αλλά πώς θα το διαχειριστούμε ακριβώς, να μην σπαταληθεί. Είναι σημαντικό να βρούμε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για να μπορέσουν ερευνητικέ ομάδες να γίνουν εταιρείε, αλλά υπάρχει ένα λεπτό όριο εκεί και γι' αυτό πιστεύω πως οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα και την ανάπτυξή τους θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες για όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Κύριο κύριος Γκρούντλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Γενικέ, ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Θέλω να σας θέσω μια ιδιαίτερη ερώτηση που σχετίζεται με το διάστημα. Στις 28 ε, ε, Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλησε να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, φορέα, διαστημικό φορέα, να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στο διάστημα, αλλά και να αναγνωρίσει το διάστημα ως καταλήτη για μια ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική. Ερώτησή μου είναι απλή. Στο επίπεδο του Horizon Ευρώπη μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι μεγάλες προτεραιότητες που έχετε εσείς διαπιστώσει να ισχύουν για αυτό το τομέα. Μπορείτε να μας πείτε ποιο ποιος προϋπολογισμός θα αφιερωθεί στο διάστημα ή εν πάση περιπτώσει ποιε είναι οι προσδοκίες σας σε αυτό το επίπεδο εφόσον υπάρχουν επίγουσες ανάγκες αυτή τη στιγμή για επενδύσεις στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα και τέλος αν μπορείτε να μας δώσετε τον τρόπο εφαρμογής ε, πώς το έχετε φανταστεί γιατί εσείς και εμείς είμαστε υπεπισμένοι για το στρατηγικό ενδιαφέρον του διαστήματος ε, στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης και του μέλλοντος της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Πακή για τις ε, εξήγησεις σας. Είπατε ότι η επιστημονική έρευνα ουσιαστικά θα πρέπει να αυξήσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι σημαντικό και συμφωνώ και άλλοι πολιτικοί κλάδοι που βάζουν πολλά χρήματα στην ε, επιστημονική έρευνα να συντονιστούν με τον ορίζοντα 2000, ε, με τον ορίζοντα. Είμαι λοιπόν στην Επιτροπή Ρέντι και πρέπει να σας πω ότι κοιτάμε και την ETC και την ε, οδηγία Interreg και έχουμε συζητήσει πολύ αυτό το παράγοντα υπαριθμών 5 σε ό,τι αφορά δηλαδή το Ταμείο το οποίο θα απλοποιήσει τον την οδό από την επιστημονική έρευνα στην υλοποίηση των προϊόντων. Υπάρχει λοιπόν κάποιος συντονιστικός ρόλος των υπευθύνων του ορίζοντα για το Ταμείο Αυτό Συμπεριλαμβάνεται αυτό στα προγράμματά σας, στο σχέδιό σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάης. Όχι δεν θέλει το λόγο, ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πακέ, υπάρχουν διάφορες ε, ε, δυνατότητες εταιρική σχέσης και ξέρετε ότι με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Ε, κυκλοφορούν διάφορα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το εξή Πώς, έχετε κάποια κριτήρια, κάποιους κανόνες για να αποφασίσετε ποιος και θα είναι ο εταίρος και έπειτα τι θα γίνει με το JTI για το διάστημα, θα, γίνει, θα υπάρξει και εταιρική σχέση ή όχι. Θέλω σαφή απάντηση. Ο κύριος Κρασνοδιεύσκη. Ναι. Ο κύριος Μαρινέσκου ήδη έθεσε αυτά τα ερωτήματα και εμένα με ενδιαφέρουν οι εταιρικέ σχέσεις. Πώς ε, και αν έχετε καταλήξει σε έναν κατάλογο, ποιο θα είναι το πρότυπο για αυτές και έπειτα αν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το ε, χρηματοδότηση των εταιρικών ε, σχέσεων. Ο κύριος Γιάμπς. Ευχαριστώ. Κύριε Πακέ, εγώ θεωρώ ότι αυτό το νέο είδος ε, συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι συναρπαστικό γιατί είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο project που θα επηρεάσει σίγουρα την ανταγωνιστικότητα ε, της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Τενοτομία, αλλά έχω δύο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σε σχέση με το στρατηγικό σχεδιασμό και τη σχετική διαδικασία, σε ποιο βαθμό η κινητικότητα του ερευνητικού προσωπικού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Παϊκό σύστημα καινοτομία και έρευνα παίζει ρόλο γιατί ε, είναι θέμα βιωσιμότητα ε, του συστήματος Ευρωπαϊκής Έρευνας και Καινοτομίας για το μέλλον, γιατί ανταγωνιζόμαστε όχι μόνο μεταξύ μας, ανάμεσα στις χώρες, ξέρουμε για το κενό της καινοτομίας λοιπά, αλλά και με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα και ίσως και άλλους ε, παίχτες. Ε, έπειτα αναφέρομαι στη συζήτηση για, που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με αυτή τη διαφορά ανάμεσα στην συνοχή και το ορίζον Ευρώπη, αν θέλετε. Δηλαδή, πού θα πάνε τα λεφτά. Αυτή η διαφορά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολύ παραγωγική και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβανόταν στο θέμα της διεύρυνσης. Πού πάνε αυτά τα χρήματα της διεύρυνσης, ε, είναι κομμάτι των τριών πυλώνων, είναι κάτι άλλο. Και έπειτα εσείς και η Κομισιόν τι πιστεύετε ε, για πιθανές συνεργασία ανάμεσα στα χρήματα της συνοχής και το ορίζοντα Ευρώπης. Είναι ε, συζητήσεις για το πώς αναφέρουν τα αποτελέσματα οι ερευνητές, ας πούμε, τα πορίσματα τους. Αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση των εθνικών σημείων επαφής. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τη γνώμη σας ποια είναι η προτίμηση της Επιτροπής σε σχέση με αυτό. Σας ευχαριστώ. Μου χρωστάτε ένα λεπτό κύριε Γιάπς. Έχω άλλους δύο ομιλητές. Την κυρία Βόντινγκ πρώτα και μετά την κυρία Τέ. Και την κυρία Γκάλβες. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γενικέ που ήρθατε ε, σήμερα να μας μιλήσετε. Πραγματικά με εντυπωσιάζει η φιλοδοξία των όσων μας προτείνατε και καλωσορίζω το γεγονός ότι αυτή η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές που θα βασίζονται περισσότερο σε ε, πορίσματα, σε αποδείξεις, σε στοιχεία. Ως ε, φιλελεύθερη είμαι εδώ για να κάνω εξατία κατά του Brexit και γι' αυτό θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τον Brexit. Ο Κάρλος Μαέδας πρόσφατα ε, σχολίασε ότι μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ένωσης και άρα έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα θέματα τα ερευνητικά και τα προγράμματα ερευνητικά όπως το Horizon 2020. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα έξι πρώτα βρετανικά ε, πανεπιστήμια ηγούνται ή συμμετέχουν σε προγράμματα ε, που ανέρχονται σε ποσά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα γίνει το Brexit. Δεν είναι αναπόφευκτο. Άρα λοιπόν, αν συμβεί, ακόμα και αν δεν το δέχομαι εγώ, τι θα γίνει με αυτά τα project, τι θα γίνει με τις ομάδες που εργάζονται από αυτών των προγραμμάτων. Δεύτερο ερώτημα, κάποιες, ε, κάποιοι διαγωνισμοί εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί και παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί το Brexit, α, εξετάζονται οι βρετανικές αιτήσει επί ίσης ώρες με τις υπόλοιπες ομάδες. Τέλος, πρόσφατη ενημέρωση για την έρευνα περί αποθήκευσης ενέργειας με τρόμο άκουσα ότι μόνο το 3% του, της έρευνας ε, που χρηματοδοτήθηκε από το Horizon 2020 σε τον τομέα ε, ήταν επιτυχές. Ξέρω πως το 100% στην έρευνα ποτέ δεν, επιτυχάνεται, αλλά το 3% είναι τρομακτικό και προφανώς υπήρξαν ε, προβλήματα από την πλευρά της της, των ερευνητών, αλλά ίσως και ήταν κακή επιλογή. Τι θα κάνετε ώστε να βελτιώσετε τα ποσοστά επιτυχίας των προγραμμάτων του Horizon Ευρώπη. Παρακαλώ όμως όταν λέω ένα λεπτό είναι ένα λεπτό ο χρόνος αγόρευσής σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την προσήλασή σας για την καταπολέμηση του καρκίνου. Όμως πραγματικά επιτυχής στατικική θα πρέπει να περιλαμβάνει και να βασίζεται επί της πολιτικής ισχύω των κρατών μελών. Εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία, όπου οι στατιστικές περί καρκίνου διαρκώς αυξάνονται. Ωστόσο, η κυβέρνησή μας δεν θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση στην ε, υγειονομική φροντίδα. Ε, εσείς προτίθεστε να συνεργαστείτε ε, με άλλα ευρωπαϊκά μέσα, όπως ας πούμε τα μέσα συνοχής, ώστε να εργαστείτε για την απόδοση, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που εσείς θα θα επιτύχετε στον ερευνητικό τομέα και αν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαψη για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων σας. Θα ήθελα πραγματικά να συμβεί αυτό και στην Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τέλος η κυρία Γκάλβες. Καταρχάς σας ευχαριστώ που ήρθατε και συγχαρητήρια. Νομίζω πως είναι εξαιρετική στρατηγική η υιοθέτηση του συστήματος των αποστολών στο πλαίσιο του Horizon Ευρώπη. Βέβαια, αυτό, η επιτυχία αυτών θα εξαρτηθεί από την ε, συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιστημών. Ε, το σύστημα των αποστολών είναι καλό όσον αφορά την κάλυψη των ανισοτήτων. Ε, εσείς προτίθεστε να κάνετε κάποιες δράσεις ώστε να πιέσετε τα κατημέλη να προχωρήσουν προς περισσότερο διεπιστημονικά συστήματα για να εκμεταλλευτούν καλύτερα το ε, σύστημα των αποστολών, γιατί διαφορετικά οι ανισότητες μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι τώρα. Ευχαριστώ. Σας υποσχέθηκα ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και μεγάλο ενδιαφέρον στο ζήτημα γενικά. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ και για το ενδιαφέρον σας και τις ερωτήσεις σας οι οποίες και δείχνουν τόσο το ενδιαφέρον όσο και τη δέσμευση της Επιτροπής. Θέλω να επιβεβαιώσω την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας, κυρία Καρβάλιο, κύριε Νίκα, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ προσωπικά, οι ομάδες μου, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρου της νέας Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομία, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή όσο εσείς θεωρείτε χρήσιμο. Σε ομάδες εργασίας πιστεύω ότι ο τρόπος είναι κάτι που θα σχεδιάσουμε μαζί. Θέλω όμως να σας επιβεβαιώσω για το γεγονός ότι είμαστε διαθέσιμοι ούτω ώστε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γνώση σας, τις επαφές σας με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε, να εμπλουτίσουμε τα στρατηγικά μας σχέδια. Στους επόμενους έξι μήνες υπάρχει χώρος για να τα κάνουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να υιοθετήθηκαν κάποια σχέδια σχετικά με κάποια Ινστιτούτα πολύ νωρί, επομένω υπάρχει χώρος και χρόνος. Πολλοί από εσά και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το, υπο, να το υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν εκρεμείς υποθέσεις, διατάξεις που δεν συζητήθηκαν μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρομαι βεβαίως σε ε, διεθνείς σχέσεις, σε ό,τι αφορά τις συνεργίες, τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αυτό βεβαίως αφορά και τις διαπραγματεύσεις για το PDP. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Απλά θέλω να ε, σας πω ότι είναι ίσως πολύ σχετικό και για μέλη που ίσως το θέλουν, να υπογραμμίσουμε την προστιθέμενη αξία του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Το άλλο βέβαια σημείο έχει να κάνει με την έρευνα. την ε, καλύτερη δυνατή επιστημονική έρευνα, προγράμματα που όχι μόνο προσελκύουν ερευνητές στην Ευρώπη, αλλά και στηρίζουν αυτούς που υπάρχουν, τους ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην επιστημονική έρευνα. Και σε όλα αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να προσθέσουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μέσω των αποστολών και των εταιρικών σχέσεών μας, ότι η έρευνα και η καινοτομία στηρίζεται σε ολόκληρο το πρόγραμμα και στη συνέχεια μπορεί να προσφέρει πολύ συγκεκριμένες λύσεις, ε, καινοτόμες λύσεις για την καθημερινότητα και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μετάβασης, την κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αλλά και για τη νέα Επίτροπο. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπογραμμιστούν ως κεντρικά στοιχεία όλα αυτά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό. Αρκετοί από εσά αναφερθήκατε στις συνεργίες. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα Horizon Ευρώπης από μόνο του δεν είναι έρευνα και καινοτομία. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να το χωρέσουμε τόσο σε εθνικό επίπεδο, οι μεγαλύτερες χορηγήσεις γίνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά από την άλλη να υπάρξουν ενεργείες και σε ολόκληρο το φάσμα του PDP να ενεργοποιηθούν είτε, είτε με τη μορφή περιφερειακών χορηγήσεων, είτε με τη μορφή πολιτιστικών πολιτικών. Σε όλα τα προγράμματα θα πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών με την ανάπτυξή τους θα ενωθούν, να δώσουμε προτεραιότητα, να προετοιμάσουμε έρευνες, να έχουμε πολλές συζητήσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλάνο το ανέφερα και στην αρχική μου παρουσίαση. Ο τρόπος που ετοιμάζουμε το πρόγραμμα αυτό είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που προετοιμάσαμε το Horizon 2020. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο ήταν εξίσου δυναμικό ας αποτελούνταν από πολλά υποπρογράμματα Υπήρχαν τα προγράμματα για την τεχνολογία, υπήρχαν τα προγράμματα για την καινοτομία, για την κινητικότητα, για την ενέργεια, για τη γεωργία, ε, τα οποία λάμβαναν χώρα σε διαφορετικά τμήματα. Βεβαίως υπήρξε ένα συντονισμός, αλλά ανήκαν ε, στην ε, εποπτεία διαφορών τμήματων. Αυτό που αποφασίσαμε όμως είναι ότι δεν θα οργανώσουμε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα αυτό, που σημαίνει ότι η Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση Connect, η Γενική Διεύθυνση Agri, η Γενική Διεύθυνση Move. Δεν έχουμε εμεί ω Επιτροπή μέρο του προπολογισμού. Κάτι το οποίο μα υποχρεώνει, αλλά και μα επιτρέπει να συνδημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τι προτεραιότητε και τη μελλοντική εφαρμογή του. Είναι μια τελείω διαφορετική προσέγγιση, το οποίο έχει αλλάξει τελείω τα δεδομένα ήδη από τον τελευταίο χρόνο και μα δίνει όθηση για περισσότερε συνεργίε από το βασιζόμενοι βεβαίως και στα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος. Μας επιτρέπει βεβαίως να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και στις διάφορες προκλήσεις τα ζητήματα δημόσιας πολιτικής. Ελπίζουμε ότι είναι σαφές το στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό είναι που ευελπιστούμε να επιτύχουμε το συνσχεδιασμό με την υποστήριξη βεβαίω του Συμβουλίου και των κρατών μελών αλλά και το, του Ευρωκοινοβουλίου. Να σας πω ότι έχω πλήρη συνείδηση ότι οι συνεργείς έχουν να κάνουν με την νομοθεσία και πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η νομοθεσία σε ό,τι αφορά α, την τεχνολογία είναι επιτάπητος. Υπάρχουν σημεία που θα πρέπει να διασαφινιστούν, να ολοκληρωθούν. Αυτή είναι δουλειά που γίνεται σε τεχνικό επίπεδο. Πέρα από αυτό όμως, οι κανονισμοί που θα επιτρέψουν όλε αυτές τις συνεργίες, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Και εδώ θα πρέπει αυτή η καινούρια προσέγγιση της Επιτροπής να το επιτρέψει. Ούτω ώστε να μπορέσουμε από κοινού να σχεδιάσουμε προγράμματα, όχι μόνο την νομοθεσία. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός στο στρατηγικό πλάνο είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Ε, δύο λόγια μόνο για τη διάσταση αυτή διεύρυνσης. Είναι ένας ε, μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού. είναι μεγάλη επιτυχία μας. Η Επιτροπή ήδη είχε προτείνει να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός. Επομένως, είμαστε σε ένα καλό ποσοστό, 3,1%. Ξέρετε ποια είναι τα σημεία που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Ένα νέο σχήμα έχει προστεθεί. για, συγκεκριμένα, για συγκεκριμένες ομάδες. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο βήμα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή. Το πακέτο διεύρυνσης όμως αυτό από μόνο του δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από ολόκληρη την Ευρώπη να σας πω ότι το πρώτο βήμα είναι η διαφάνεια του στρατηγικού σχεδιασμού. Τίποτα δεν γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Όλα τα Ινστιτούτα, όλα τα πανεπιστήμια γνωρίζουν, είναι, ε, είναι προσκεκλημένα να συμμετάσχουν. Τώρα λοιπόν ε, διοργανώνουμε την εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως υπάρχει και ευθύνη που έχει να κάνει με τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο επικοινωνίας σε κάθε κράτος και τα κράτη, το καθένα από αυτά θα πρέπει να είναι ενεργό σε όλη αυτή τη διαδικασία, να μπορέσει να συμμετάσχει, ούτω ώστε να προετοιμαστούν για την καλύτερη εφαρμογή. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι όλη αυτή η ανοιχτή Δικασία προετοιμασίας του προγράμματος δημιουργεί και μια πιο ευέλικτη βάση. Ανοίγει το δρόμο για πολύ, περισσότερο, για πολύ περισσότερες ε, διαβουλεύσεις, σε πολύ περισσότερα τμήματα, ε, κοινωνικές επιστήμες, υψηλά, χαμηλά τεχνικά επίπεδα. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Όλοι οι τομείς αυτής, σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουμε... Ε, ενδιαφερόμενα μέρη που δουλεύουν μαζί μας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καλή κάλυψη, μια πολύ μεγαλύτερη ευρία εφαρμογή του ορίζον Ευρώπη. Η επιτυχία μας είναι κυρίως επιτυχία στην επιλογή σε μερικές ε, περιπτώσεις έχουμε μια χαμηλή, ένα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ε, διαπιστώσει στις συζητήσεις μας και καθώς προετοιμάζουμε την εφαρμογή συζητάμε για προτεραιότητες πολιτικής. Θα περάσουμε πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει καλή κατανόηση Γίνονται επίσης έρευνες αξιολόγησης, εκθέσεις αξιολόγησης για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουμε βελτιωθεί και για να έχουμε και καλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο μέλλον. Υπήρξαν κάποια σχόλια και για το Brexit. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι φορτισμένο πολιτικό, πολιτικά είναι ιδιαίτερα καμφώδες. Να σας πω ότι όδο σήμερα επισήμως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως συμμετάσχει στο πρόγραμμα που συζητάμε και στην εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει μέρος του προγράμματος. Μέχρι να ολοκληρωθεί τουλάχιστον το Horizon 2020. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει τρίτη χώρα, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το κάθε project κατά περίπτωση. Να δούμε πώς συμμετέχουν ως μεμονωμένα μέλη. Ένα σενάριο no deal είναι ένα σενάριο που θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια διαφορετική έκβαση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις μας, η έρευνα και η καινοτομία είναι ένας τομέας που είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως πολύ σημαντικός Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εργαστεί πάνω στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αρκετοί από σας είπατε ότι υπάρχουν διατάξεις στην πρόταση της Επιτροπής που θα πρέπει να συζητηθούν στο Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά βιομηχανικές τρίτες χώρες με ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα. Αυτό θα είναι μια δυνατότητα που υπάρχει στο, στο πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Δεν υπήρχε στο Horizon 2020. Ε, αυτό είναι σημαντικό για τις μελλοντικέ σχέσεις με τρίτες χώρες. Προς το παρόν όμως επικεντρωνόμαστε στις επόμενες εβδομάδες. Είναι σημαντικό να πούμε δύο λόγια η διερμηνία θα τελειώσει. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, λοιπόν. Ε, σε ό,τι αφορά την στόχου για το νορίζοντα 2020, ελπίζουμε να βελτιωθούν οι συνθήκες μέχρι το τέλος του 2020 για την εφαρμογή. Δεν προγραμματίζουμε λοιπόν συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα τα οποία στην ουσία να είναι διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, αλλά από την άλλη είναι πολύ διαφορετικό το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί ο ορίζοντας Ευρώπης. Ξέρετε ότι για την υποψήφια πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, μια πράσινη συμφωνία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Και εδώ θα έχουμε βασικό ρόλο για την τεχνολογία, το κοινωνικό σκέλος της κοινοτομίας και αυτά προσπαθούμε να πετύχουμε λοιπόν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχω μεγάλες φιλοδοξίες και το Κοινοβουλίο επίση σε ό,τι αφορά την διάσταση του κλίματος για το μελλοντικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει προφανώς ανταγωνισμός μεταξύ EIT και EIC. Έγιναν πολλές συζητήσεις μεταξύ διαφόρων φορέων και το Ευρωπαϊκό ε, Ινστιτούτο για Τεχνολογία είναι βασικό σκέλος στο τρίγωνο της ε, γνώσης στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την ε, γνώση και σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Αυτό θα συνεχίσουμε να το προωθούμε και τουλάχιστον αυτό κάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι η επιπλέον αξία σε ό,τι αφορά το EIT και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πλέον ε, εμπλέκεται στην στρατηγική, στο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν το κοιτάμε ξεχωριστά. Και έτσι να δούμε και το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το οποίο θα μπορεί να λεφθεί υπόψη πλήρω πλέον και να εφαρμόζονται είτε από το EIC, είτε από άλλα μέρη του προγράμματος. Άρα φαντάζομαι ότι μεταξύ EIC, EIT, μεταξύ των ε, ε, πάνελ, μεταξύ όλων των φορέων θα είναι πιο ομαλή. Έτσι εργαζόμαστε από αυτόν στο, στο, στην Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά το EIT, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EIC σε άλλες ε, υπηρεσίες. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίε. δυσκολίες, δεν υπάρχουν δυσκολίες. Τώρα ποια θα είναι η επόμενη φάση, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, ούτε θέλω να το σχολιάσω. Και πρόεδρε, να πω ότι οι περιοχές με έντονη κατανάλωση άνθρακα, όλα αυτά έχουν εντοπιστεί στις διαπραγματεύσεις, αποτυπώνονται στις διαπραγματεύσεις, θα υποστηρίξουμε λοιπόν την μετάβασή τους και αυτό παραμένει προτεραιότητα για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για τις ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να απαντήσω, θα μπορέσω να τις απαντήσω κατά, κατηδίαν. Και ξέχασα για το διάστημα να μιλήσω. Μου επιτρέπετε. Για το διάστημα, προφανώς αποτελεί προτεραιότητα για την ε, υπηρεσία μας και στη φάση της διαπραγμάτευσης το διάστημα ε, μπήκε στο ψηφιακό σκέλος και στο σκέλος ε, το σκέλος του διαστήματος και προφανώς η χρηματοδότηση για το διάστημα είναι τμήμα της χρηματοδοτικής αλλά και της στρατηγικής του στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε λοιπόν όμως μόνο σε αυτό το σκέλος γιατί προφανώς το διάστημα αποτελεί μια υπηρεσία και για τις μεταφορές, για την γεωργία, για την ασφάλεια, για την υγεία Άρα η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός προφανώς ε, έχουν να κάνουν και με άλλα σκέλη του προγράμματος και προφανώς ε, έχουν να κάνουν και με τη φιλοδοξία που έχει αποφασιστεί μεταξύ της Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου αλλά και πολλών άλλων για την πρόθεση των εφαρμογών του διαστήματος σε περίπτωση και μια συνεργασία για το διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαρινέσκου, που θα συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Γενική Δευθυντά, για το χρόνο που μας αφιερώσατε, για τις απαντήσεις σας. Και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μόνο η απαρχή της διαδικασίας. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό και θα ακούσουμε όλο και πιο πολλά. Θα ακούμε όλο και πιο πολλές πληροφορίες από το Γενικό Διευθυντή και από τους υπόλοιπους. Τα λέμε λοιπόν πάλι στις 2.30. Λήξη της συνεδρίασης.